Ε, good morning, colleagues. Καλημέρα σας συνάδελφοι. Ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην ημερήσια διάταξη, αλλαγές τελευταίας στιγμής. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, για τις σχέσεις με την Αραβική ε, χερσόνησο για την αποστολή στη Σαουδική Αραβία. Ο κύριος Καν δεν είναι σε θέση να έρθει σήμερα να μας μιλήσει. Θα τον δούμε λοιπόν στις 26 Μαρτίου. Ο Ρίτσαρτ Χάουιτ που σκόπευε να μας παρουσιάσει έκθεση από το Φόρουμ των Ηνωμένων Αθηνών για τις επιχειρήσεις και τις σχέσεις με τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει, ανα... έχει ματαιώσει αυτήν την ε, ε, παρουσίαση γιατί χρειάζονται επαφές με την κοινότητα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα πρέπει να συζητήσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με τις ε, ε, με τις, ε, με τις σκληρές ποινές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές κυρώσεις. Αυτό αναβάλλεται. Βλέπω ότι σημειώνεται τις αλλαγές μας στην ημερήσια διάταξη και στην έγκριση των πρακτικών της 5ης Φεβρουαρίου, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Τα εγκρίνουμε. Ανακοινώσεις λοιπόν. Ξεκινώ με, τα, με τις καλές ειδήσει σε σχέση με το Καζακστάν. Το έχουμε συστήσει και στην υποεπιτροπή μας έχει αποφασίσει ο Υπουργό των Εξωτερικών της Ισπανίας να απορρίψει το αίτημα για έκδοση του κυρίου Μουράτμπεκ και που είχε υποβάλει το Καζακστάν. Απόφαση που θεωρούμε πολύ θετική, την είχαμε ζητήσει εξάλλου και επανειλημμένως είχαμε ζητήσει από το Προεδρείο την απόρριψη του αιτήματος για έκδοση. Σε σχέση δε με τον κύριο Μουκτάρ Αμπλιάτσοφ. Έχουμε αποστείλει αντίστοιχα επισκευή, επιστολή στον στο Γαλλικό Υπουργείο των Εξωτερικών για την ε, αίτηση έκδοσης εις βάρος του. Ελπίζουμε ότι και ο Γάλλος Υπουργός των Εξωτερικών θα βρει το θάρρος, όπως ε, επέδειξε ο Ισπανός Υπουργός, να απορρίψει ε, αυτό το αίτημα. Για το Στρασβούργο είχαμε πολλά θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην προηγούμενη σύνοδο. Την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο για το 2013 και την πολιτική της Ένωσης στα θέματα αυτά με πολύ καλά αποτελέσματα στις προφορίες της έκθεσης Παντσιέρη. Κάποιες από τις συστάσεις είναι πολύ σημαντικές για τη δουλειά μας. Λέμε παραδείγματι ότι θα πρέπει να υπερασπίσει περισσότερο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους αγωνιστές των δικαιωμάτων που βρίσκονται στη φυλακή και θα πρέπει να υπάρχει μια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που να παρακολουθεί την κατάσταση στην συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών σε περίπτωση που έχουμε κρατουμένους αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε δε στην ημερήσια μας διάταξη για σήμερα μια ανταλλαγή ε, απόψεων με τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης ζητούμε την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών για τις διακοινοβουλευτικέ αντιπροσωπείες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία του Κοινοβουλίου και ζητούμε οι κατευθυντήριες γραμμές να ακολουθούνται από, να συζητηθούν από την διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών σε συνεργασία με την, Επιτροπή, με υποεπιτροπή μας. Επίσης το ψήφισμα ενθαρρύνουμε να, να προαχθούν οι συζητήσεις ε, για την ενσωμάτωση των διαφορών μέσων που έχει διαθεσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προαγωγή και την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα στρατηγικό έγγραφο. Μια μικρή φράση που σημαίνει πάρα πολύ δουλειά. Εάν χρειαστεί να το κάνουμε αυτό, εάν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, θα έχουμε πάρα πολύ δουλειά στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γιατί θα πρέπει να ηγηθούμε της σύνταξης μιας της στρατηγικής. Μετά έχουμε το, είχαμε το ψήφισμα του ε, ηγέτη της αντιπολίτευσης Μπορίς Νεμτσόφ και τα θέματα τα σχετικά με τη δημοκρατία στη Ρωσία, όπου καταδικάστηκε η δολοφονία του Νέμτσοφ και η περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης των δικαιωμάτων στη Ρωσία. Ε, επικρίνουμε επίσης νέες διατάξεις που εισήχθησαν προκειμένου να περιοριστεί η δράση της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών και την κράτηση της ε, Νάντια Σαυτσέγκο, του Αλέκτσεϊ Ναβάλνη και του Όλεκ Ναβάλνη. Καταγγέλουμε επίσης τον πόλεμο κατά των θεμελιωδών και δημοκρατικών αξιών. Είχαμε επίση ε, ψήφισμα για την κατάσταση του Νότιο Σουδάν και ιδιαίτερα εκφράσαμε τις ανησυχίε μας στα θέματα της ασφάλειας, στα ανθρωπιστικά θέματα στο Νότιο Σουδάν που θα μπορούσαν να προξενήσουν αποσταθεροποίηση σε ολόκληρη την ε, περιοχή της νοτιοανατολικής ε, της Βορειοανατολικής Αφρικής και καλούμε σε κατάπαυση πυρός άμεση και πλήρη και ασφαλή επάνωδο των παιδιών που έχουν απαχθεί από τις ένοπλες δυνάμεις, από τις αρχές της ένοπλης σύγκρουσης το 2013. Κατεπήγον είχαμε επίσης σε σχέση με τους φετερισμούς γεών στην Τανζανία. Με, το για, με την πρόθεση μάλλον ε, ανακοινωθήσα πρόθεση για πώληση 1.500 τετραγωνικών χιλιόμετρων στην περιοχή των Μασάι προκειμένου να απολυθεί αυτή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για λόγους διεξαγωγής αφάρι και κυνηγιού. αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εκδιωχθούν από τις γέες του 40.000 βοσκοί Μασάι. Ζητούμε να πάψει αυτό και να γίνει διερεύνηση των διαφορών έγκυας ιδιοκτησίας στην περιοχή Λολιόντο. Και μετά είχαμε τις πρόσφατες επιθέσεις κατά των ε, σύρων χριστιανών και τα εγκλήματα του λεγόμενου Ικίλ. Είχαμε αυτή τη συζήτηση, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον επίσκοπο, τον σύρο επίσκοπο από τον Λίβανο, αλλά και εκπρόσωπο της Συριακής Κοινότητας του Ιράκ στην επίσκεψη αυτή ε, όταν πήγαμε. Θερμά μας ευχαρίστησαν για το ψήφισμά μας και η κατάσταση στη χώρα είναι κρίσιμη. Προσπαθούν να ε, φυγαδεύσουν χριστιανούς Σύρους στον Λίβανο για να τους σώσουν. Ξέρουμε ότι τα ψηφίσματά μας μπορεί να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά πάντως είναι παρήγορο το ότι μπορούν να βοηθούν τους ανθρώπους αυτούς. Επίσης σημειώνουμε στο ψήφισμα αυτό ότι δεν μπορεί να νοηθεί ατιμορρησία για τους αυτούργους αυτών των εγκλημάτων, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, εγκλημάτων πολέμου και ότι θα πρέπει να παραπεμφθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η κυρία Σούντι ο επικεφαλής αγγελέας είχε ήδη ανακοινώσει τη σχετική πρόθεση για παραπομπή τέτοιων πολεμιστών όταν προέρχονται από χώρες που έχουν κυρώσει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Μετά έχουμε τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνδέσμου Αραβικών Κρατών και συνεργασία στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Έχουμε ε, ζητήσει να κοινοποιούνται τα πρακτικά των εργασιών του συνδέσμου. Έχουμε ζητήσει από τα αραβικά κράτη να σέβονται την απαγόρευση των βασανιστήριων όπως τα γνωρίζει η Σύμβαση για την απαγόρευση των βασανιστήριων. Βλέπω ότι ίσως να σας κουράζω, αλλά έχουμε πολλά ψηφίσματα στα ανθρώπινα δικαιώματα από την προηγούμενη σύνοδο. Έχουμε ακόμα ένα για τη Βενεζουέλα, όπου ζητούμε ελεύθερη και ανοιχτή συζήτηση μεταξύ κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως. Καλούμε με το ψήφισμα την κυβέρνηση να κάνει σεβαστό το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας και κάθε διεθνή σύμβαση και συνθήκη που έχει προσυπογράψει η Βενεζουέλα. Στο ψήφισμα καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς ε, τις ε, δικαστικές έρευνες και δίκες που λαμβάνουν χώρα στη χώρα και εν τέλει είχαμε το ψήφισμα για τις προτεραιότητες για το 2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της 28ης Συνόδου του Συμβουλίου των Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Αύριο θα έχουμε την αποστολή μας στην Γενέβη που θα ε, στηριχθεί στο ψήφισμα αυτό για τις συζητήσεις του Συμβουλίου με τους διπλωμάτες εκεί. Με τα λύπης μου σημειώνω πάντως ότι το ψήφισμα υιοθετήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ώστε να ληφθεί ε, δεν, μπορεί να είναι, δεν μπόρεσε να είναι καιρός έτοιμο ώστε να ληφθεί υπόψη από την Ολομέλεια όταν θα έρθει η ώρα. Και προτείνω άλλη φορά να ετοιμαζόμαστε πολύ ταχύτερα, πολύ νωρίτερα. Αυτά. Βλέπετε νομίζω και εσείς σε ποιου τομεί εργαζόμαστε. Αυτό είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Η Επιτροπή μας είναι κομμάτι τη ε, της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων. Ασχολούμαστε με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι εντός. Αυτό είναι δουλειά άλλη Επιτροπής. Και χαιρόμαστε που σα έχουμε εσάς εδώ για να μας παρουσιάσετε ως ειδικό την κατάσταση στην Ερυθρέα. Η κυρία Σίρα Κίταροτ, λοιπόν, η ειδική εκπρόσωπος από τα ανθρώπινα δικαιώματα της στην Ερυθρέα και μέλος της Επιτροπής Έρευνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθρέα, θα μας ε, παρουσιάσει δε η Επιτροπή σας ε, τα πορίσματά της τον Ιούνιο του 2015 στο Συμβουλίο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και βλέπω στα χαρτιά μου, στρέφομαι εδώ και προς εσάς, εσείς να μας βοηθήσετε, ε, ότι έχουμε προσκαλέσει και τον κύριο Άντεν Μπραν Βέλτε Τζόρτζης. Μάλιστα, έχει κολλήσει όμως την κίνηση και έρχεται. Είναι πρώην πρέσβης της Ερυθρέας στο Βέλγιο. Έχει δημοσιεύσει μάλιστα και βιβλίο η Ερυθρέα ως σταυροδρόμη. Θα τον ακούσουμε όμως όταν έρθει. Προσκαλέσαμε ή προσπαθήσαμε να προσκαλέσουμε και εκπρόσωπο της πρεσβείας της Ερυθρέας. Αλλά δεν κατέστη δυνατό να λάβουμε απάντηση θετική και συμμετοχή στην Επιτροπή μας. Είμαι βεβαία ότι οτιδήποτε συζητούμε εδώ φτάνει πάντα στις πρεσβείες, στον πολιτικό. Φαντάζομαι ότι και η Ερυθρέα θα ενημερωθεί. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Ας ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε εσείς. Και όταν έρθει ο κύριος Βέλτε Τζόρτζης, τον ακούμε ή ιδάλλως ξεκινούμε τη συζήτηση. Κυρία του παρακαλώ. Good morning, ladies and gentlemen. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εξοχότητες. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας ενημερώσω για την Ερυθρέα. Γιατί πιστεύω ότι είναι καθήκον μου να σας ενημερώσω ε, για θέματα της Ερυθρέας ε, και γενικώ να ε, εκμεταλλεύομαι κάθε ευκαιρία και να εμφανίζομαι σε πολλά φόρα προκειμένου να γύρω το θέμα της Ερυθρέας. Θα σας κάνω μια σύντομη εισαγωγή και να σας ε, αναφέρω το ιστορικό της εντολής του ειδικού εισηγητού για την Ερυθρέα. Θα σας αναφέρω την προσέγγιση μου, να σας ε, πω δύο λόγια για το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής και να σας ε, μιλήσω εν συντομία για τους πρόσφυγες και τους ετώντες άσυλο από την Ερυθρέα. Από, πού προσπαθούν, από τι προσπαθούν να ξεφύγουν αυτοί οι άνθρωποι, τι προσπαθούν να γλιτώσουν και επίσης κάποια καταληκτικά σχόλια και συμπεράσματα. Καταρχήν για το έργο μου. Η εντολή αυτή δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2012. Δεν πρόκειται να διαβάσω ολόκληρο το ψήφισμα 2020 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Πάντως, η εντολή δημιουργήθηκε εξαιτία τη βαθύτατη ανησυχία των συνεχών κατάφορων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τι αρχέ τη Ερυθρέα εις βάρος του πληθυσμού της Ερυθρέας και των επικών ε, με παραβίαση πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών δικαιωμάτων και δεδομένου του ανησυχητικού αριθμού ε, πολιτών της Ερυθρέας που προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα εξαιτία των κατάφορων αυτών παραβιάσεων. Αυτό προβλέπει το ψήφισμα 2020 του Συμβουλίου Ασφαλείας του, του Συμβουλίου, Ασφαλείας για τα, του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ. Συνεχίζω. Την ίδια περίπου εποχή το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέτασε την κατάσταση ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα σε κεκλεισμένο των θυρών ε, συνεδριάσεις, ε, κρατώντας τον εμπιστευτικό χαρακτήρα στην ανάλυση κάποιων ειδικών υποθέσεων και ζήτησε από την κυβέρνηση Ερυθρέας να παράσχει πληροφορίες στην 21η Σύνοδο που έλαβε χώρα τον ε, Σεπτέμβριο του 2012. Και όταν ε, δημιουργήθηκε αυτή η εντολή και η θητεία του ειδικού εισηγητού, συνέβη κάτι πρωτοφανές για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δηλαδή, αυτές οι απόρριτες ε, υποθέσεις δημοσιεύθηκαν με κάποιες ε, διορθώσεις ε, από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επιδόθηκαν στον ειδικό εισηγητή για συνέχιση της εξέτασης και της εξυχνίασης αυτών των υποθέσεων. Αυτά λοιπόν είναι τα καθήκοντά μου γέννη. Βέβαια, ως θα φαντάζεστε. Η απάντηση της Ερυθρέας ε, είναι ότι η εντολή αυτή έχει πολιτικά κίνητρα, ότι δεν συνάδει με τις ε, ειδικέ εντολές αναχώρα και ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο εξαιτίας της καθολικής περιοδικής ε, εξέτασης που κάνει επαρκή αξιολόγηση των, της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μέλων του ΟΗΕ και γι' αυτό δεν έχω καμία πρόσβαση στην επικράτεια της Ερυθρέας. Είχαμε πέρυσι το δεύτερο γύρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκδόθηκαν 200 περίπου συστάσεις, γιατί στον πρώτο γύρο συστάσεων δεν είχαμε τη δέουσα εφαρμογή. Για το δεύτερο γύρο συστάσεων είχαμε μια επιλεκτική αποδοχή κατά τη γνώμη μου, 90 συστάσεων από τις 200. Οπότε η καθολική περιοδική εξέταση είναι μια καλή διαδικασία, αλλά η απάντηση χώρα είναι σχετικά χαλαρή. Και αν δούμε τις επιδόσεις της χώρας ό,τι αφορά την καθολική περιοδική εξέταση, σε σχέση με τον πρώτο και τον δεύτερο γύρο, βλέπουμε τις διαφορές. Βέβαια, η Ερυθρέα μας ενημέρωσε ότι έχει συστήσει μια επιτροπή για να εξετάσει τη συμμόρφωση των συστάσεων της καθολικής περιοδικής εξέτασης, του UPR. Τώρα, όταν δημιουργήθηκε αυτή η εντολή για τη θητεία μου, εγώ εξέτασα ποια είναι, τι κάνει ο ειδικό ηγετή σε τέτοιε χώρε, ποια είναι τα καθήκοντά του. Και έπεσε σε μία δήλωση πρώην ειδικού εισηγητή που λέει ότι εμείς θέτουμε την προστασία των Αρχόντων ανάγκη ως προτεραιότητα και υιοθετούμε μία προσέγγιση που προσανατολίζεται στο θύμα, στα θύματα. Αναλύουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προβαίνουμε σε συστάσεις και πασχίζουμε να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη ε, υπέρ των θυμάτων, των πραγματικών και των ανθρώπων που υφίστανται απειλέ. Ασθενίζουμε αυτή την προσέγγιση και γι' αυτό προσπάθησα να διαμορφώσω και τη δική μου προσέγγιση. Η εντολή ε, επιτρέπει εξέταση κατάσταση στην Ερυθρέα προκειμένου να βρεθούν αηφόρες ε, βιώσιμες λύσεις ε, που θα πληρούν τις προδιαγραφές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι κάτι που επισημαίνω συνεχώς στις αρμόδιες αρχές της Ερυθρέας. Επαναλαμβάνω όμως ότι η κυβέρνηση της Ερυθρέας απέρριψε ευθύ εξ αρχή την εντολή του ειδικού εισηγητού του ΟΗΕ για τη χώρα αυτή, οπότε δεν έγιναν καν συζητήσεις. Η προσέγγιση μου είναι συγκρατημένα αισιόδοξη. Ε, θέλω να εφαρμόσω στα έπακρα την εντολή, να επικεντρωθώ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα και να δώσω φωνή σε χιλιάδες κατοίκους Ερυθρέας που πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα να υψώσουν τη φωνή τους. Ε, ήρθε σε επαφή μαζί τους ε, σε επισκέψεις μου σε άλλες χώρες και η ανανέωση της εντολής της εντολής μου θα εξεταστεί το 2015. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ειδική Εξεταστική Επιτροπή που συστήθηκε πέρυσι, έργο της θα είναι η διερεύνηση, παρόλο που και αυτή η Επιτροπή απορρίφθηκε από τις αρχές της Ερυθρέας, η τελική έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής θα υποβληθεί τον Ιούνιο χθε μάλιστα είχαμε μια προφορική ενημέρωση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε το τελευταίο τμήμα. Αυτό που είπε ο Πρόεδρος είναι ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η μαζική έξοδος ε, κατοίκων της Ερυθρέας ε, δεν μπορεί και δεν θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί χωρίς ε, να αντιμετωπίσουμε προηγουμένως την ανθρωπιστική κατάσταση, κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Αυτό είναι το επίκεντρο της συζήτησης, η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάποια αριθμητικά στοιχεία, εντάχει, χωρίς λεπτομέρειες, γιατί σας έχουμε δώσει λεπτομεριακά στοιχεία. Αυτά ήταν τα στοιχεία που έλαβα και εγώ όταν ξεκίνησα τον διαδραστικό διάλογο με την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών πέρυσι. 4.000 το μήνα περίπου. Βέβαια έχουμε σκαμπανεβάσματα, αλλά 4.000 είναι ο μέσος όρος. 4.000 άνθρωποι το μήνα. Αλλά υπάρχει μια μικρή αύξηση που θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Η καταστροφή τραγωδία της Λαμπεντούζα είναι γνωστή σε όλους. Δεν χρειάζεται να σταθώ σε αυτήν. Ήταν πάντως μια τραγωδία που δεν θα πρέπει να λησμονηθεί. Τώρα, τι είπε ένας από τους ε, συνομιλητές μου. Τι γίνεται όταν κάνει... Τι γνώμη έχει να μείνει κανείς στην Ερυθρέα όταν δεν μπορεί να βοηθήσει τους οικείους του όταν ε, είναι αναγκασμένος να λάβει κάποιες αποφάσεις, να διακινδυνεύσει τη ζωή του είτε στην έρημο είτε ε, διασχίζοντας τη θάλασσα, γιατί είναι απελπισμένος. Και ελάχιστες είναι οι ελπίδες του. Ακόμη και να ε, τα καταφέρει, ακόμη όταν είναι κανείς στο σκοτάδι, ακόμη και μία ακτίδα φωτός ε, δίνει την ελπίδα και την, ε, το θάρρος να αναλάβει κανείς ένα τέτοιο κίνδυνο. Νομίζω ότι αυτό είναι ενδεικτικό της κατάστασης ε, που επικρατεί στην Ερυθρέα και που είναι συνειφασμένη και με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κατάλογος είναι μακροσκελής, μπορείτε να διαβάσετε τις εκθέσεις μου έχουμε την, ε, την ε, στρατιωτική θητεία και οι παραβιάσεις που γίνονται στα πλαίσια της ε, υπηρεσίας αυτής της στρατιωτικής θητείας. έχει σχέση και με τη διάρκεια της θητείας. Επίσης, σεξουαλική κακοποίηση των γυναικών, εξοδικαστικές συνοπτικές εκτελέσεις, αναγκαστικές εξαφανίσεις. Είναι μερικές περιπτώσεις παραβίας ανθρωπινών δικαιωμάτων. Πάντως ε, είδαμε από τα προηγούμενα σχόλια την απόγνωση όσων ε, προσπαθούν να γλιτώσουν από την Ερυθρέα που αναλαμβάνουν τον κίνδυνο αυτού του πολύ επικίνδυνου ταξιδιού προκειμένου να ξεφύγουν από τη χώρα. Ξέρω ότι υπερεύει το χρόνο μου. Θα ήθελα απλώς να συμπληρώσω ότι πιστεύω και να επαναλάβω εδώ την έκκληση μου προς τη διεθνή κοινότητα ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενισχύσει τις προσπάθειές της ε, για να αποτραπεί, να αποφευχθεί η επανάληψη της τραγωδίας της Λαμπεντούσα. Και να λάβουμε υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό συνόδευτων ανηλίκων ε, που φεύγουν από την Ερυθρέα και από συζητήσεις που είχα σε καταβλισμούς ε, προσφύγων διαπιστώνω ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός να, γίνει σεβαστή αυτή η αρχή της και να δοθεί, αν όχι άσυλο, τουλάχιστον προσωρινό κατάλημα σε όσους το χρειάζονται. Είναι θεμελιώδου σημασία επίσης το γεγονός ότι διμερείς και άλλες συμφωνίες μεταξύ της Ερυθρέας και τρίτων χωρών που διακυβεύουν ε, τη ή υπονομεύουν ε, την ε, ζωή όσων ζητούν άσυλο θα πρέπει να σταματήσουν. Επίσης υπάρχει και ελαθρεμπόριο και παράνομη διακίνηση. Αλλά αυτά τα φαινόμενα της διακίνησης και της σωματεμπορίας είναι απλώς συμπτώματα, είναι κρούσματα συγκεκριμένων ειδικών προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έσωθεν και κυρίως να χτυπηθούν τα αίτια του κακού και οι λόγοι που εξωθούν αυτούς τους ανθρώπους στη φυγή από την πατρίδα τους. Αυτά και είμαι έτοιμη για συζήτηση. Σας ευχαριστώ κυρία Κίταρουτ. Ήταν πολύ πυκνά το όσα μας εξηγήσατε και τώρα προχωρούμε. Μας πει ο κύριος Άντερμαντ Τζόρτζες, που είναι ο πρέσβης στο Βέλγιο της Ερυθρέας και γράψει επίσης και ένα βιβλίο «Η Ερυθρέα σε Σταυροδρόμι». Μια αφήγηση θριάμβου και ελπίδας. Μπορείτε να μας κάνετε μια εισήγηση ένα δεκάλεπτο και κατόπιν να συζητήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα. Συγγνώμη που καθυστέρησα να φτάσω, αλλά έμπλεξα στην ε, κίνηση. Ερχόμουν από το Βατερλό. Είχα προγραμματίσει να έρθω εδώ 8 και 4 και έλεγα τι θα κάνω μέχρι τις 9 ε, και τελικά έφτασα μια ώρα αργότερα από τις 8 και Τέλος πάντων, πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω την κυρία Ελένα Βαλεντιάνο και γενικότερα την Υποεπιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου γιατί ε, οργάνωσε αυτή τη συνάντηση και με καλέσατε για να συμμετάσχω και να ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα. Επίσης, για να δω και εσάς κυρία, μια πολύ ευχάριστη στιγμή να είμαστε εδώ μαζί για να συζητούμε τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πατρίδα μου και πάρα πολύ συχνά δυσκολεύεται κανείς να πιστέψει ότι η κατάσταση των δικαιωμάτων είναι τόσο άσχημη σε μια χώρα. Σε μια χώρα η οποία αναδύθηκε από τις τάχτες ενός ε, τόσο μακρού, μακροχρόνιου πολέμου πριν από 25 χρόνια, γιατί έχουμε όλες αυτές τις ιστορίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθρέα. Και Ακριβώς είναι αυτέ οι ιστορίες πολύ, πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς. Είχαμε αυτόν τον πόλεμο, γίνανε θυσίε για ελευθερία, ευημερία, δικαιοσύνη και το 1991 είχαμε την ε, απελευθέρωση για μια καινούργια αρχή τη χώρα, αισιοδοξία, ελπίδα για μια καλύτερη ζωή για τον λαό της χώρας. Δυστυχώς όμως αυτή η χαραυγή, αυτή η Ανατολή τελικά έγινε Δύση, έγινε σούρουπο, έγινε μία νύχτα και τις ε, λεπτομέρειες τις ε, ακούσατε, τις, τις εξήγησε τόσο καλά η δική εκπρόσωπος. Καταλήξαμε στο ανάποδο αυτού για το οποίο πολεμήσαμε. Το γιατί είναι μια μεγάλη ιστορία. Όλα αυτά προσπάθησα να τα περιγράψω στο βιβλίο που έγραψα. Σήμερα θέλω να κεντρώσω την προσοχή μου πρώτα-πρώτα στην απουσία του κράτους δικαίου. Δεύτερον, στο ότι έχουν ακυρωθεί, έχουν ενεργηθεί βασικές ελευθερίες. Τρίτον, παραβίαση των δικαιωμάτων και να κλείσουμε με ένα τέταρτο σημείο. Κάποιες προτάσεις για το τι μπορεί να γίνει ούτω ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και γενικότερα στη χώρα μου. Πρώτα-πρώτα, ανθρώπινα δικαιώματα. Το Σύνταγμα της χώρας, μεταξύ άλλων, ορίζει την, τον τρόπο λειτουργίας, την αρμόδια αρχή της λειτουργίας και επίσης οριοθετεί τη, το, το μέχρι που φτάνουν οι τρεις βασικές εξουσίες. Η επιτελεστική, Επίση περιγράφονται τα βασικά δικαιώματα οπότε απαιτείται από το κράτος να τα περιορίσει και ως νομικό θεμέλιο του κράτους έχουμε την εθνική κυριαρχία και επίσης πηγή κάθε νομιμότητα είναι η, το, το, το κοινοβούλιο σύμφωνα με το σύνταγμα το σύνταγμα αυτό εγκρίθηκε το 97 στο τέλος μιας μεγάλης μεταβατικής ε, περίοδου. Και με αυτό το σύνταγμα θα είχαμε δημοκρατία και επίσης έτσι θα είχαμε την άσκηση της διακυβέρνησης με βάση του κράτους δικαίου. Θα ισχύουν σήμερα. Όμως έχει κλείσει από το 2001 αυτή η Βουλή. Η ιδέα δικαστική εξουσία υφίσταται συνεχείς παρεμβάσεις από την εκτελεστική εξουσία. Υπάρχει η Προεδρία της χώρας που κυριαρχεί στην ζωή της χώρας, την πολιτική και κοινωνική. Και τελικά ο κρατικός μηχανισμός έχει κατασταλτική λειτουργία. Οπότε ο λαός μας υφίσταται συνεχή παραβίαση των δικαιωμάτων τους, των ελευθεριών, της αξιοπρέπειας και δεν έχουν ε, κάποιο καταφύγιο, κάποιο τρόπο διαμαρτυρίας. Μιλάμε για τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες. Δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης του... Ε, πώς του συνέρχεστε ή του συνεταιρίζεστε. Και η εθνική ασφάλεια καταστέλει έκφραση απόψεων της αντιπολίτευσης, κάποιοι επίκριση κατά την κυβέρνηση, όλα αυτά έχουν ποινικοποιηθεί. Και επομένως υπάρχει πάρα πολύ αυστηρός έλεγχος, οπότε όπως ε, εξήγησε η ειδική εισηγητής, αν τον κόσμο να φύγει. Γι' αυτό και βλέπουμε επίσης ε, πάρα πολύ κόσμο να περιμένει να φάνε το δελτίο, πάρα πολλούς να έχουν ε, όπλα ή τόσο πολλοί ζουν στις γειτονικές χώρες σε κάποια άθλια στρατόπεδα ε, επίσης βλέπουμε πτώματα ακροτηριασμένα και θα έχετε δει όλες αυτές τις φρικτές εικόνες είδαμε πόσοι πνίγονται στην Μεσόγειο, όπως έγινε στην ε, Λαμπεντούζα, την Ιταλική νήσο. Επίσης έχουμε αυτή την βίαιη καταστολή, πάρα πολύ φτώχεια. Κατεδάφιση σπιτιών στην πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις και κατάσταση επιδεινούνται συνέχεια. Να, τι κυριαρχεί στην σημερινή Ερυθρέα. Για να δούμε τι γίνεται με την παραβίαση των δικαιωμάτων. Έχουμε κάποιες προσπάθειες να προβληθούν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά η απάντηση είναι συλλήψεις, φυλάκιση και βασανισμοί. Οπότε βλέπουμε πώς καταστρέφεται η ζωή του κόσμου, πώς διαλύονται οι οικογένειες και πώς έχει ανασταλεί η λειτουργία της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει δίκαιη δίκη. Ούτε απαγγέλλεται καμία κατηγορία και με ισχυρισμού κατηγορίες, υποψίες είναι κάτι το οποίο αρχίζει να μπει κανεί στη φυλακή χωρί να υπάρχει για όποιον τα υποστεί αυτά καμία βοήθεια. Οπότε δεν υπάρχει το δικαίωμα τη υπεράσπισης, ε, δεν έχει επαφή με τον έξω κόσμο και επίση δεν επιτρέπεται να τον επισκεφθούν οι φίλοι, η οικογένεια και αντίθετα με τη βασική νομική αρχή του τεκμήρου της αθωότητας εκεί ισχύει το αντίστροφο. Μέσα στο τοποθετεί κάτι αντίστοιχο θεωρείται ότι είναι ένοχος και παραμένει σε κράτηση. Οπότε βλέπετε τι γίνεται και με την υγεία όλων αυτών των φραγισμένων και διαφόρων ε, ε, υπαλλήλων του προηγούμενου καθεστώτος, δημοσιογράφων και απλών πολιτών οι οποίοι κρατούνται και σε απομόνωση από το 2011. Τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, η διεθνή κοινότητα. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα θα πρέπει να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση. Ούτω ώστε να πιστεί η κυβέρνηση να υλοποιήσει, να εφαρμόσει το Σύνταγμα, να εφαρμόσει το κράτος δικαίου. Δεύτερον, κάτι θα πρέπει να γίνει με αυτές τις αυθαίρετες συλλήψεις, τις επάρους των ε, κρατήσεις, τα βασανιστήρια και τις ε, εκτελέσεις χωρίς δικαστική απόφαση. Να απελευθερωθούν όλοι αυτοί οι πολιτικοί οι κρατούμενοι, οι απλοί άνθρωποι, οι δημοσιογράφοι κλπ. Τέταρτον, θα πρέπει να δούμε ε, να υπάρξει κανονική στατολόγηση και να σταματήσουν στατολογούν τους νέους. Επίσης, να υπάρχει υποχρέωση ε, λογοδοσίας για τα οικονομικά και σωστή κατανομή των πόρων σύμφωνα με τα όσα σχήνει διεθνώς. Επίσης, έβδομο και πάρα πολύ σημαντικό, οι διεθνείς κοινότητες και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσουν στις προσπάθειές μας και στην Ερυθρία αλλά και από πλευράς διασποράς τόσο ώστε να υπάρξει μία μετάβαση σε δημοκρατικό καθεστώς. Για να δούμε τι, τι, γίνεται με τα χρόνια δικαιώματα για να δει κανείς τι ισχύει γενικά στη χώρα σας παραπέμπω στο βιβλίο μου το οποίο το παρουσιάσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Παρασκευή. Να το, βιβλίο εδώ το κρατώ. Και σας είπα ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό γιατί λέμε ε, ότι εκεί δεν έχουμε ελευθερία συνεταιρίζεστε, ελευθερία έκφρασης, συναθρίζεστε και, και επομένως δεν μπορούμε να συζητήσουμε ποιο θα είναι το μέλλον της χώρας τι αλλαγή θα πρέπει να γίνει, τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν. Ούτε υπάρχουν κάποιοι θεσμικοί μηχανισμοί για διαδοχή στην ηγεσία της χώρας, ο αντιπρόεδρος κλπ. Επομένως θα έχουμε κενό εξουσίας το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αιματοχυσία και χάος. πρέπει να αποφύγουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Γι' αυτό και θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσουν την υποστήριξή τους για να γίνει αυτό ο δημοκρατικός μετασχηματισμός στη χώρα μας και σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βέλντε Τζόρτζες. Πολύ συγκεκριμένη η τοποθέτηση και η περιγραφή σας. Είπατε ότι θα πρέπει να ασκηθούν αποτελεσματικές πιέσεις στην κυβέρνηση της Ερυθρέας. Πώς όμως θα γίνει αυτό. Θα ακούσουμε τώρα, εάν θέλει, να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση, η κυρία Μπράουν ή η κυρία Κορέα είναι εδώ. Καλημέρα σας. Και καταρχάς ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρουσιάσεις, για την παρουσίαση της κυρίας Κίταρουτ ως προς την κατάσταση των δικαιωμάτων στην Ερυθρία και ευχαριστώ και εσάς κύριε Πρέσβη. Εν γέννηση μεριζόμαστε τις ε, θέση σας. Βλέπουμε όμως ότι έχει κάνει σημαντικά βήματα, έστω και πολύ μικρά η Ερυθρέα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, εμείς καλωσορίζουμε και υποστηρίζουμε το διάλογο με την Ερυθρέα, γιατί θεωρούμε ότι ο διάλογος είναι ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλιστεί, ελπίζουμε, πρόοδος εν γέννη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, λοιπόν, στο διάλογο με την Ερυθρέα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μια προσέγγιση με βάση σαφείς αρχές. Επιμένουμε δηλαδή στο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα Μας απασχολεί η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων στην Ερυθρέα. Ένα ζήτημα το οποίο σε κάθε ευκαιρία που προσφέρεται γύρουμε. Είχαμε παραδείγματι τον κύριο Γιμάνι Γκεμπρέμ, τον κύριο σύμβουλο του Πρωθυπουργού μαζί με τον Υπουργό των Εξωτερικών που επισκέφθησαν τις Βρυξέλλες πρόσφατα. Ε, σε αυτούς θέσαμε το ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων. Τους επισημάναμε ότι, έχουμε, ότι πρέπει να γίνει κάτι, ότι, έχουμε, ότι υπάρχουν κρατούμενοι από το 2001. Ο κύριος Ισακτάβιτ επίσης, ο Έλμαρ Μπρόκ, ο ευρωβουλευτής που υποδέχθηκε την ίδια την προσωπία, επέμεινε στο θέμα αυτό, είπε ότι έχει πια έρθει η ώρα να αποφυλακιστούν οι κρατούμενοι αυτοί από το 2001. Δεν έχει πια κανένα νόημα να παραμένουν στη φυλακή. Είναι βαρύτατη η παραδοτών Η κράτηση των ανθρώπων αυτών χωρίς δίκη. Σταματώ εδώ προς το παρόν. Αλλά θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό να ε, αναπτύσσουμε και να διατηρούμε το διάλογο με την Ερυθρέα και να πιέζουμε για γενική ε, πρόοδο. Έχουμε εντατικές επαφές και κονδύλια που έχουν προβλεφθεί για την Ερυθρέα με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Θέλω επίση να υπογραμμίσω σε σχέση με τους πολιτικούς κρατουμένους ότι είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται κάθε φορά, πατή εκπρόσωπος των εξωτερικών, μάλλον εκπρόσωπος της υπάτης εκπροσώπου, κάθε χρόνο δημοσιεύει δήλωση με την οποία καλείται η κυβέρνηση της Ερυθρέας να αποφυλακίσει τους πολιτικούς κρατουμένους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Λόχπιλερ. Ο κύριος Αντακ... Αντάκτουσον. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Περιμένω να βάλετε ακουστικά σας. Tack så mycket. Eh, alla vi som har arbetat med... Eh, ευχαριστώ. Όσοι εξημών έχουν ε, ασχοληθεί με την Ερυθρέα και τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί, ξέρουμε πολύ καλά ότι επικρατεί ένα σκληρό καθεστώς, ένα καθεστώ το οποίο πολύ εύκολα μετέρχεται βία για να εξυπηρετήσει τους στόχους του. Εγώ έχω ασχοληθεί με τα θέματα της Ερυθρέας εδώ και χρόνια. Παρακολουθώ την ε, κατάσταση σχέση με τον ε, Derek Ισακ που προέρχεται από τη Σουηδία όπως και εγώ ε, και είναι κρατούμενος. Έχουμε πολλούς Ερυθρέους επίσης στη Σουηδία και μπορώ να παρακολουθώ την κατάσταση μέσω αυτών. Με ενισχύει ιδιαίτερα λοιπόν σχέση με τους πολιτικούς κρατουμένους το εξή. ότι το καθεστώς φαίνεται απολύτως αδιάφορο σε οποιαδήποτε προσπάθεια για άσκηση πολιτικών πιέσεων, είτε από την Σουηδική κυβέρνηση, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εστιαστώ λοιπόν σε ένα ερώτημα που επανέρχεται στις συζητήσεις με τους εξόριστους Ερυθρέους και αφορά την φορολογία του 2% που επιβάλλει το καθεστώς της Ερυθρέας στους ε, ομογενείς ή εξόριστους Ερυθρέους που ζουν στο εξωτερικό που αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματο για το καθεστώ. Εμά στη Σουηδία μα έχει αποσχολήσει πολύ αυτό. Θέλουμε να δούμε δηλαδή αν αυτό το ποσό του φόρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πίεσης. Παρακολουθώ λοιπόν τις συζητήσεις και ρωτώ εάν μπορείτε να απαντήσετε μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό σε ένα μέσο πολιτικής πίεσης προς το καθεστώς, εάν πούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν δεχόμαστε, ότι δεν δέχονται αυτό το είδος ε, φορολογίας, αυτό το φόρο. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το συνδυάσουμε και με το Συμβούλιο Ασφαλείας που λέει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι πολιτικές. Μήπως αυτό μπορεί να, ασκηθεί, να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης για την αποφυλάκηση των πολιτικών κρατουμένων. Η κυρία Βεργιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχουμε επιτέλους την ευκαιρία να συζητήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθρέα. Ευχαριστώ τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών που μας βοηθάει. Χωρίς την έκθεση σας νομίζω δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τη σημερινή συζήτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Και όπως πραγματυπώθηκε η Ερυθρέα είναι η μία από τις χειρότερες δικτατορίες του κόσμου, αν όχι η χειρότερη θα επικεντρωθώ σε δύο-τρία παραδείγματα. Στην διεθνή κατάταξη στη χειρότερη θέση έχει 6.000 πολιτικούς κρατουμένους για 6 εκατομμύρια ε, κατοίκους, νούμερο αντίστοιχο με αυτό της Τουρκίας, που χωρίς να θέλω να πω ότι χαίρομαι που έχουν τόσους κρατουμένους στην Τουρκία, εν πάση περιπτώσει είναι πολύ μεγαλύτερη χώρα ε, απόλυτη λογοκρισία από το 2001 στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν υπάρχει δυνατότητα έκφρασης άλλης από αυτήν που υποδεικνύει η κυβέρνηση. Ε, σύνταγμα που υφίσταται εδώ και πολύ καιρό δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή εθνικές εκλογές, βουλευτικές εκλογές από το 1993 αναβάλλονται διαρκώς, δεν έχουν γίνει εκλογές από το 1993 στην Ερυθρία, κανενός είδους εκλογική αναμέτρηση. Πιστεύω λοιπόν ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουμε, μείνει, έχουμε ε, βρεθεί να υπολοιπόμεθα των περιστάσεων. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εγείρουν τη φωνή του για την παραμικρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένε χώρε, ενώ για την Ερυθρέα σιωπούμε. Και πολλές φορές απολύτω. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω να γίνεται συζήτηση δε, για τέτοιο θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο. Ένα ψήφισμα το 2011, ένα από τα ελάχιστα ψηφίσματα που αφορούσα ε, ειδικά την κατάσταση του κυρίου Νταβί Βιζάκ, Σουηδο-Ερυθρέου, του οποίου παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα. Τι κάναμε λοιπόν εμείς για αυτόν τον Ευρωπαίο υπήκο, εντωμεταξύ, και άκουσα, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας δώσετε παραπάνω πληροφορίες, ότι εκφράζονταν και ανησυχίες ακόμη για τη ζωή του κύριου Νταβίζακ. Το ίμιση των κρατουμένων, των πολιτικών κρατουμένων στην Ερυθρέα έχει αποβιώσει τι είδους χώρα είναι αυτή στην οποία μπορεί να εκδηλώνεται μια τέτοια κατάσταση και εμείς να μην, στην, να μην αντιδρούμε. Ακούω να μιλάει η Επιτροπή και με άφωνη. Με συγχωρείτε κυρία μου, δεν εννοώ εσάς προσωπικά, τη δουλειά σας κάνετε. Αλλά όταν μας λέτε μικρά μικρά βήματα στα ανθρώπινα δικαιώματα, επίτε μας λοιπόν, σας κλιπαρώ, ποια βήματα έχουν πραγματοποιηθεί. Και όταν λέτε εσείς ότι κοφεύει το καθεστώς. Ε, τι πολιτικό διάλογο μπορούμε να αναπτύξουμε με μια χώρα που κοφεύει και αδιαφορεί απολύτως για οτιδήποτε έχουμε να πούμε, άσε που δεν λέμε και τίποτα. Τι κάνουμε, τι, ποια είναι τα τελευταία εφευρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διάλογο που αναπτύσσει με την Ερυθρέα, διαδικασία του χαρτούμ. Το είπατε συγκεκαλυμμένα εσείς, κυρία Κίταρουτ. Είπατε θα διαπραγματευτούμε με τις κυβερνήσεις των χωρών του κέρατος Αφρικής για το θέμα των μεταναστών. Μα αυτούς που προσπαθούν να ξεφύγουν από καθεστώτα κατασταλτικά και αφόρητα, τι θα διαπραγματευτούμε για τα θέματα, για τους ανθρώπους αυτούς, τι θα επιτύχουμε. Και θα συμφωνήσω με αυτό που υπόθηκε νωρίτερα. Ένα όπλο είναι τα κονδύλια η Ερυθρέα είναι κράτος που έχει συνυπογράψει τη συμφωνία του Κοτονού. Τη συμφωνία του Κοτονού. Ε, πρέπει λοιπόν να ενεργοποιηθούν οι ρήτρε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν σε χώρα όπω η Ερυθρέα δεν εφαρμόζεται αυτέ, πού πάμε, πού πορευόμαστε, τι είμαστε, βάση περιπτώσει. Και επιπλέον, όλοι αυτοί οι Ερυθρέοι που ζουν έξω από τη χώρα, χωρί τη χρηματοδότησή του αυτών των ομογενών, δεν θα είχε σταθεί το καθεστώς. Οι ίδιοι οι επιτρέπουν την επιβίωση όσων δεν μπορούν να ξεφύγουν σε τελευταία ανάλυση με, τις, με, ε, με τα εμβάσματά τους. Ε, πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε διαφορετικά τη χώρα αυτή. Είναι αφόρητο να έχουμε φτάσει στην ίδια κατάσταση και να μην παρακολουθούμε τακτικά τις εξελίξεις. Ελπίζω η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών να μας δώσει τη σχετική ευκαιρία και παρακαλώ να παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή την κατάσταση του Νταβίν Ιζακ, γιατί πρόκειται για μια υποδειγματική περίπτωση, πρόκειται για μια περίπτωση με την οποία μπορούμε και να κινητοποιήσουμε και την κοινή γνώμη να εξηγήσουμε το τι συμβαίνει. Και πάνω απ' όλα πρέπει να εξασφαλίσουμε, να βεβαιωθούμε ότι ζει ακόμη. Και εν τέλει, από αυτά που είπατε, και νομίζω συμφωνούν με τα όσα καταγράφει στην έκθεση του τους εκπρόσωπους για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο θέμα των προσφύγων. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την χορήγηση διεθνούς προστασίας σε όποιους τη χρειάζονται και κυρίως τους ανηλίκους. Κυρία Λόχπίλερ. Ο κύριος Αυστρεβίτσιος έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας που μας ενημέρωσαν για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Και η σημερινή συζήτηση θα ξαναφέρει στο επίκεντρο την Ερυθρέα και την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελπίζω να επανερχόμαστε στο θέμα αυτό τακτικά και στο μέλλον. Κυρία Κίταρουτ, έχω δύο ερωτήσεις. Μια και δεν έχετε πρόσβαση στην επικράτεια της Ερυθρέας, ε, δεν είστε ευπρόσδεκτοι από τις αρχές και σας έχει εμποδιστεί η στη χώρα αυτή. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τι είδους ανταλλαγές απόψεων έχετε με αυτούς ε, τους εκπροσώπους και τι κάνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, έχουν δράσει στην Ερυθρέα. Η διεθνή κοινότητα έχει, το δικό της, έχει στείλει το δικό της μήνυμα προς τις αρχές της Ερυθρέας. Ρωτώ λοιπόν, αυτό το μήνυμα φτάνει στην κοινωνία των πολιτών της χώρας αυτής. Γιατί από ό,τι μας είπατε, οι αρχές ελέγχουν πλήρως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την επικοινωνία και τη ροή πληροφοριών. Οπότε οι ντόπιοι έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητη πληροφόρηση από άλλες πηγές, έχουν, μπορούν να ακούν σταθμούς ε, από άλλες χώρες ή να ενημερώνονται. Μας είπατε ότι έχει αυξηθεί η μεταναστευτική ροή από την Ερυθρέα. Σε ποιο βαθμό αυτές οι μεταναστευτικές ροές οφείλονται σε πολιτικούς ή οικονομικούς λόγους γιατί μια και η οικονομία της Ερυθρέας βρίσκεται σε δίνη κατάσταση και μια και δεν υπάρχει ούτε οικονομική ούτε κοινωνική ανάπτυξη στη χώρα, μπορεί τα κίνητρα της μετανάστευσης να μην είναι μόνο πολιτικά, αλλά να είναι και οικονομικά. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για το ποια είναι τα πραγματικά αίτια της μετανάστευσης ή τουλάχιστον των πρόσφατων μεταναστευτικών ροών από την Ερυθρέα. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ. Ευχαριστώ αν δεν κάνω λάθος, ε, γύρω στο 2000... Ε, είμαι 16 χρόνια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη μοναδική συζήτηση που είχαμε ε, τότε για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα είχα λάβει το λόγο και θυμάμαι ότι τότε είχα ζητήσει να ανασταλεί η Συμφωνία του Κοτονού. Γιατί ακόμη και τότε είχε ήδη 10 χρόνια κυβέρνηση από το 1991 και δημιουργήθηκε ένα, διδακτορικό καθεστώς, ένα δικτατορικό καθεστώς και ένα βασίλειο του τρόμου. Και νομίζω ότι η Ερυθρέα είναι η Βόρεια Κορέα της Αφρικής. Και μάλιστα στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, στην έκθεσή μου για το κέρας της Αφρικής, Είχα συζητήσει με τον ειδικό εκπρόσωπο για το κέρα τη Αφρική και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπήρχε η αίσθηση ότι από τη στιγμή που δεν μπορούσαμε να αναστείλουμε την συμφωνία του Κοτονού, έπρεπε να κρατήσουμε την αντιπροσωπεία μα στην Ασμάρα, την πρωτεύουσα τη Ερυθρέα, για να κρατήσουμε ε, ένα είδο πίεση στο καθεστώ. Δεν έχω όμω την αίσθηση ότι ασκήσαμε κάποια πίεση, γιατί έχει ε, επιδεινωθεί η κατάσταση και δεν ξέρω αν 120 εκατομμύρια αναπτυξιακή βοήθεια ε, έχει νόημα να ε, στέλνονται προς αυτή την κατεύθυνση, μια και δεν υπάρχουν καθόλου βελτιώσει ό,τι αφορά το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι λυπηρή η κατάσταση και άθλια η μέχρι στιγμής ιστορία της Ερυθρέας. Είχαμε την, τον πόλεμο με την Αιθιοπία, τη μαζική επιστράτευση νέων, διαλυμένη οικονομία. Δεν έχει μείνει ουσιαστικά ε, κανένας Ερυθρέος. Οι μισοί είναι στις φυλακές. Ε, είναι ένα αποσταθρωμένο κράτος. Ε, ο δικτάτορας ελέγχει κάθε μορφή της πολιτικής και της οικονομίας. Έχω όμως ένα διαφορετικό σχόλιο. Πριν από μερικά χρόνια ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ο πρόεδρος φαίνεται να χρηματοδοτεί τρομοκρατικές ομάδες στην Αφρική και ιδιαίτερα στη Σομαλία γιατί ο εχθρός του εχθρού σου είναι φίλος σου και θεωρήθηκε ότι θα μπορούσαν να ήταν εχθροί της Αιθιοπίας. Ισχύει εμπάργο όπλων προς την Ερυθρέα ή μπορεί ακόμη να χρηματοδοτεί το δικτατορικό καθεστώς ε, τρομοκρατικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Μία σύντομη ερώτηση προς την εκπρόσωπο της ΕΙΕΔ. Και θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με τη διαδικασία του Χαρτούμ για την Ερυθρέα. Και συνεχίζεται ο διάλογος με την κυβέρνηση. Και αν ε, ζητάτε στα πλαίσια αυτού του διαλόγου να εξασφαλιστεί πρόσβαση της ειδική ηγήτριας του ΟΗΕ στη χώρα αυτή. Όπως μας υπενθύμησε ο κύριος Στάνοκ, δεν υπάρχει καμία πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε, αντί αυτή την περιπτώση, γιατί να μην ε, ανασταλεί η συμμετοχή τη Ερυθρέας από τη Συμφωνία του Κοτονού. Πολλές ερωτήσει, ε, αλλά αυτό το νόημα έχει συζήτηση. Λοιπόν, ξεκινούμε από την ειδική συγγετρία του ΙΕ. Ευχαριστώ πολύ, ειδική συγκεντρία. Πρώτα απ' όλα για αυτό το φόρο του 2% μέσω πολιτική πίεσης, τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να θεωρηθεί η κατάσταση, γιατί πάρα πολύ ξεκάθαρα εξηγείται το τι γίνεται στα πλαίσια των κυρώσεων εις βάρος τη Ερυθρέας. Δεν είμαι ειδική στο θέμα, αλλά τέλος πάντων ενημερώνομαι. Και έχουμε κάποια παραδείγματα ε, χωρών που εφαρμόζουν τέτοιο φόρο. Ο Καναδάς και πρόσφατα το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε σχετικές καταγγελίες από ε, ε, κατοίκους σε σχέση με αυτό. Τώρα τι μπορεί να γίνει. Ακριβώ γιατί υπάρχουν παραδείγματα για περιστατικά του να επιβαρύνονται με αυτό το 2%. Και υπάρχει ποικιλία αντιδράσεων από χώρα σε χώρα. Στα γαλλικά συμφωνώ 100% όσον αφορά τους πολιτικούς κρατουμένους κλπ. Έχετε δίκιο. Ισχύει αυτό το οποίο είπατε. Επίσης ε, δεν ξέρω τι, πώς, πώς παρακολουθείτε το θέμα από τη δική σου οπτική γωνία, αλλά που είναι κάτι απαράδεκτο. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορούμε τώρα να επισύλλουμε στις λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ σημαντικό η υπόθεση της Ερυθρέας να παραμείνει ζωντανή στο θεματολόγιο και να συζητείτε. Επομένως, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Επίσης, για την προσβασιμότητα που είπατε, δεν υπάρχουν μη κυβερνητικέ οργανώσει που να δρούν στην Ερυθρέα. Δεν υπάρχουν αγωνιστέ για ανθρώπινα δικαιώματα οι οποίοι να βγουν να διατρανώσουν τι ε, απόψει του, να τοποθετηθούν στα διάφορα προβλήματα. Και από ό,τι γνωρίζω, υπάρχουν κάποιε αιστείε αντίσταση. Να, Φερρυπίν όταν αποφάσισαν κάποιες οικογένειες ότι δεν θα στείλουν τα παιδιά τους ε, στα κέντρα στρατολογίας. Αλλά δεν έχουμε ανεξάρτητες μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχουν κάποιες τέτοιες οργανώσεις με συγκεκριμένη γραμμή πλεύσης σε σχέση με τις κυβερνητικές πολιτικές. Είδατε για τις ε, συζητήσεις για το γυναικείο ζήτημα στη χώρα, το οποίο το, το, το κατέβασε βέβαια μια οργάνωση. Αλλά δεν έχουμε άλλες τέτοιες περιπτώσεις για συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένες ε, παραβιάσεις των δικαιωμάτων, ας πούμε σεξουαλική κακοποίηση στα πλαίσια του στρατού. Είχα επαφή με κάποιους αγωνιστές στην ανθρώπινα δικαιώματα και κάποιους ε, ε, νομικούς που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλοι αυτοί ε, όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Ε, οπότε βέβαια και τώρα με την ευκαιρία θέλω να τους ευχαριστήσω όλους εκείνους. Αλλά κανείς δεν έχει πρόσβαση σε κάποιον, πώς θα να κάνει επαφές και συζητήσεις. Οπότε και αυτοί με βοήθησαν να αναδείξω το πρόβλημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην ε, Ερυθρέα. Επομένω, για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα, ε, σύμφωνα με την έρευνα που έχω διεξαγάγει, διαπίστωσα ότι παραβιάση των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι εκείνο το οποίο ε, προκαλεί αυτήν την έξοδο όλων αυτών όπως σας εξήγησα και δεν ξέρω τώρα να το θεωρήσουμε πολιτικό οικονομικό φαινόμενο τι να σας πω ας διαπιστώσουμε ότι αν ο μόνος εργοδότης είναι η κυβέρνηση στα πλαίσια του στρατού με, τι εργασιακά δικαιώματα να έχεις τι εργασιακά δικαιώματα να ασκήσει κανείς στο ελεύθερο εμπόριο Άρα επομένω και το ζήτημα αυτό έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό από την οπτική γωνία των εργασιακών δικαιωμάτων. Εάν ο ανθός της χώρας είναι στον στρατό, τότε τι δραστηριότητα να αναπτυχθεί. Τι έχω μιλήσει σε άλλους, σε γυναίκες που έχουν ένα πάγκο και πουλάνε τσάι ας πούμε, αλλά πέραν αυτό, τι γίνεται με το δικαίωμα στην εργασία. Έτσι βλέπω εγώ τα πράγματα και θα πρέπει να θέτουμε το ερώτημα. Ο πλευρά οικονομική δραστηριότητα, τι παραβίαση δικαιωμάτων υπάρχουν και ποιες είναι οι οικονομικές συνέπειες. Οι προοπτικές δεν είναι βίωνες. Πώς να ασκήσει κανείς ένα επάγγελμα, ε, αμπόριο, Εάν κανείς δεν είναι στο στρατό, πάλι δουλεύει για το κράτος και κάνει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, σας είπα ότι όλα αυτά τα έχουμε εξετάσει και πέραν αυτών που σας είπα έχουμε και τις σχέσεις με την τρομοκρατία. Σομαλία και Ερυθρέα. Υπάρχει κάποια ομάδα που παρακολουθεί τι γίνεται. Γιατί σύμφωνα με την εντολή μου καλύπτεται και αυτή η δραστηριότητα. Είναι η εντολή που μου έδωσε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για την Κοτονού τώρα δεν έχω και πολλά στοιχεία να σας αναφέρω για ενημέρωση αλλά το θέμα είναι πώς και πού θα μιλοποιηθεί η προστασία των δικαιωμάτων για εκείνους οι οποίοι φεύγουν για να γλιτώσουν από την βίαιη ε, παραβίαση των εθνικών δικαιωμάτων. Τι να πρωτοπεί κανείς. Τόσα πολλά τα προβλήματα. Το θέμα είναι πώς θα προστατεύσουν αυτόν τον κόσμο. Γιατί ε, το θέμα είναι τι ισχύει από πλευρά διεθνού δικαίου για του πρόσφυγε. Η σα ευχαριστούμε. Έχετε το λόγο, κύριε. Μα ρωτήσατε συγκεκριμένα. Όχι απαραίτητα αλλά θα ήθελα να συμπληρώσω το είπε η κυρία Κίτερουτ. Και σε αυτά που είπε η εκπρόσωπος υπηρεσίας εξωτερικής δράσης θα ήθελα να τοποθετηθώ. Πιστεύω όντως ότι η επικοινωνία, οι συνομιλίες είναι πολύ σημαντικές αυτή η διαδικασία, είναι η μόνη προσέγγιση, αλλά όχι πάση θυσία, δεν μπορεί να είναι επικοινωνία δηλαδή σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Υπάρχουν κάποια θεμελιώδη ζητήματα, ουσιώδη του κοτονού, που μπορούμε πιστεύω να τα χρησιμοποιήσουμε ως μέσα για να επιφέρουμε άνοιγμα του οικονομικού και πολιτικού χώρου. Βέβαια η αναπτυξιακή συνεργασία με ένα καθεστώς το οποίο δεν έχει ακόμα δημόσιο προσωπολογισμό. Κανείς δεν γνωρίζει ποιες είναι οι πηγές των εσόδων του και πού πηγαίνουν οι δαπάνες του. Πρόσφατα είδαμε ταχύτατες εξελίξεις στον εξορρυκτικό τομέα, στα ορυχεία και αν δείτε τα ισοζύγια και τις δηλώσεις της κυβέρνησης βλέπουμε ότι 200 εκατομμύρια το χρόνο αντλεί η κυβέρνηση από τα ε, αξιόγραφα και από τα τέλη διαχείρισης και εξόρυξης χρυσού και αργύρου. αργύρου. 40% είναι τα διακρατούμενα, είναι το, το ποσοστό των διακρατούμενων ε, αξιών σε έσοδα για την κυβέρνηση. Το μέτωπο βασικά, έτσι, όχι η κυβέρνηση, γιατί το μέτωπο βρίσκεται μπροστά. Έτσι λοιπόν έχουμε περί τα 200 εκατομμύρια που εισπράττει η κυβέρνηση. Πού πάνε όμω τα λεφτά αυτά. Ο Υπουργό των δεν γνωρίζει, η Κεντρική Τράπεζα δεν γνωρίζει. Εγώ από ιδιωτικέ πηγέ γνωρίζω ότι βρίσκονται σε τράπεζες τη Κίνας στο όνομα ενός ατόμου. Πού πάνε τα χρήματα αυτά. Ένας φυσικός πόρος θα έπρεπε κανονικά να είναι ευλογία για μια χώρα, να αξιοποιείται για να βελτιώνεται μια κατάσταση που διαβιούν αυτοί οι άνθρωποι αυτοί που είναι φρικτοί, το γνωρίζουμε όλοι. Πώς μπορούμε λοιπόν να συνομιλήσουμε και να έχουμε επαφές με την κυβέρνηση χρησιμοποιώντας την αναπτυξιακή συνεργασία ως εργαλείο, ως μέσο μόχλευσης. Δεν θα μας πει βέβαια ότι δεν χρειάζεται την εξωτερική βοήθεια και θα πορευθεί ανεξάρτητα. Χρειάζεται λοιπόν τη μόχλευση αυτή και μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Υπάρχουν και θέματα που αφορούν την κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση ε, εκμεταλλεύεται τα προσχήματα ώστε να μετατρέπει την κατάσταση αυτή σε μια επίσημη μορφή δουλείας. Το 1994 ανακηρύχθηκε το καθεστώς Έχουμε να κάνουμε μια μικρή χώρα. Χαρήκαμε στην αρχή γιατί είναι, μικρή χώρα και δεν μπορούσε να διατηρεί μεγάλο στρατό. Και εγώ που ήμουν μέλος της Εθνοσυνέλευσης τότε θεώρησα ότι καλά πάμε με διαπεριφερειακή συνεργασία, ε, ανάπτυξη κτλ. Καλού κακού θελήσαμε να είναι εκπαιδευμένο ο λαός μας ε, με το σύστημα τη Ελβετία. Έξι μήνες εκπαίδευση στρατιωτική και ένα χρόνο δηλαδή ε, υπηρεσία κοινωνική ε, στο Σουδάν. Αυτό ήταν το σχέδιό μας. Τώρα, ένας νέος, μια νέα κοπέλα με το σύστημα που υιοθετήθηκε το 1994 έχει ξεκινήσει με το σύστημα αυτό και έχει φτάσει στα 39-40. Όλα αυτά τα χρόνια δουλεύει δωρεάν για το κράτος χωρίς να αμείβεται. Παντρεύεται, κάνει παιδιά, δεν μπορεί να, τα, να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του. Τι κάνετε λοιπόν. Αυτοί είναι οι οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες που προξενούν την ε, ε, μετανάστευση. Εγώ σας λέω ότι είναι οικονομική πάνω απ' όλα. Είναι μια δουλεία απαράδεκτη για τον 21ο αιώνα. Μη αμοιβόμενη εργασία. Όλα αυτά τα ορυχεία, Καναδί... Αυστραλοί, Κινέζοι που τα εκμεταλλεύονται. Ορυχείο, μάλιστα τώρα έχουν βρει και ορυχείο καλίου το οποίο από ό,τι ξέρω ξεπερνάει και τα μεγέθη της Ρωσίας και του Καναδά ακόμα. Στριμώχνονται ποιος θα πρωτοπιάσει, ποιος θα πρωτοβρει ευκαιρία να το εκμεταλλευτεί. Με δουλειά όμως των ε, Αιθιοπών η οποία δεν αμείβεται γιατί να πρέπει κανείς να εξαναγκάζεται στον 21ο αιώνα να δουλεύει χωρίς να αμείβεται. Γι' αυτό το λόγο φεύγουν οι άνθρωποι. Φεύγουν, εγκαταλείπουν τη χώρα, αναλαμβάνοντας ένα τεράστιο κίνδυνο, γιατί υπάρχει εντολή για τους συνοριοφύλακες να εκτελούν όποιον βλέπουν να προσπαθεί να διαβεί τα σύνορα. Στη συνέχεια έχουν να διαβούν τη Σαχάρα για να φτάσουν στα, στις όχθες της Μεσογείου αν επιβιώσουν και να προσπαθήσουν να ξεμπαρκάρουν στην Λαμπεντούσα με όλους τους κινδύνους και τις τραγωδίες που βλέπουμε συχνά. Και μετά βλέπουμε τι συμβαίνει από την άλλη μεριά στους νεαρούς Ερυθρέους του... στην περιοχή του Σινά, όπου έχουν μείνει ανεξέλεγκτα τα σύνορα όλους αυτούς τους κινδύνους είναι διατεθειμένοι οι άνθρωποι αυτοί να τους αναλάβουν, να τους διατρέξουν, προκειμένου να ξεφύγουν από μια κατάσταση αφόρητη. Αφόρητη για τους ανθρώπους αυτούς. Δεν μπορούν να ζήσουν έτσι πια στην Ερυθρία. Και αυτή είναι η πραγματικότητα που τους κάνει να εγκαταλείπουν τη χώρα τους. Όχι υποσχέσεις ή κάτι άλλο που ακούστηκε. Εγώ θα προτιμούσα να γυρίσω να ζήσω, να ζήσω στην πατρίδα μου. Δεν υπάρχει τίποτα σαν την πατρίδα αλλά κινδυνεύω να θέσω τη ζωή μου σε κίνδυνο. Όπως οι ε, προηγούμενοι σύντροφοι και συναγωνιστές, κινδυνεύω κι εγώ να χάσω τη ζωή μου. Δεν υπάρχει λοιπόν απασχόληση, δεν υπάρχει απασχόληση με κατάλληλη αμοιβή, είναι ε, στάσιμη η κυβέρνηση, η οικονομία. Η κυβέρνηση δεν ασχολείται καθόλου με μακροοικονομικές στατιστικές και δεδομένα, άρα έχουμε πολύ περιορισμένους ε, πολύ περιορισμένες πηγές που να δίνουν στατιστικά στοιχεία. Οι, οι φορείς του Bretton Woods λίγο πολύ δίνουν κάποια στοιχεία που πάντως μας δείχνουν ότι δεν είναι επαρκή τα επίπεδα διαβίωσης έξω από τη μιζαρία για του ανθρώπους αυτού. Ευχαριστώ. Και τώρα εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής δράση. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις ε, πολύ εύστοχες και περιεκτικές ερωτήσεις. Καταρχήν η θέση της ΑΕΔ σε ό,τι αφορά τη θέση του ειδικού εκπροσώπου του ΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθρία. Σας διαβεβαιώ ότι κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία, είτε στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου που έχουμε μία φορά το χρόνο με την κυβέρνηση της ε, Ερυθρέας, αλλά και στις συναντήσεις που έχουμε με μέλη της κυβέρνησης, <coughs> πάντοτε επιμένουμε στην ανάγκη να εξασφαλιστεί πρόσβαση ε, δική σας ε, στην Ερυθρέα για να δείτε ειδή σώμα στην κατάσταση και ζητούμε και πρόσβαση και στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής στην Ερυθρέα για να κάνουν το έργο της ε, και επίσης ε, πρόσβαση στον πρόεδρο της ομάδας παρακολούθησης ε, Ερυθρέας Σομαλίας. Επιμένουμε λοιπόν να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε κάθε φορά που έχουμε συναντήσει με εκπροσώπους Ερυθρέας και επιμένουμε στην ανάγκη συνεργασία της χώρας αυτής με τα Ηνωμένα Έθνη. Δεύτερον, για το θέμα της προόδου. Γιατί ανέφερα σε κάποια δηλαβήματα προόδου ε, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθρέα. Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι πέρυσι το Δεκέμβριο ο πρόεδρος της Ερυθρέας ε, ανήγγειλε μείωση, περιορισμό της στρατητικής θητείας ε, για τους νέους εφέδρους σε 18 μήνες, αντί να είναι απεριόριστη η στρατητική θητεία. Τώρα θα περιορίζεται από εδώ και πέρα στους 18 μήνες. Βέβαια είναι αργή η πρόοδος και θα συνεχίσουμε τις, τα διαβήματα. Θα ζητήσουμε μάλιστα την κυβέρνηση να, να δημοσιεύσει αυτό το μέτρο και φυσικά θα πρέπει να παρακολουθούμε εκ του και στον τρόπο εφαρμογής. Γιατί αυτή η απεριόριστη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, όπως είπατε κι εσείς, χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση φθηνού εργατικού δυναμικού. Και αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερος και μας προβληματίζει. Θα δούμε τώρα αν η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τα μέτρα που εξήγηλε για τον περιορισμό της στρατητικής θητείας. Ένα άλλο θέμα είναι ότι έχουν απελευθερωθεί 7 δημοσιογράφοι τον Ιανουάριο από τις φυλακές ε, που κρατούνταν από το 2009. Εντάξει, δεν είναι και καμιά φοβερή πρόοδος, αλλά είναι ένα μικρό βήμα. Επίσης, η κυβέρνηση προσπαθεί να εφαρμόσει τις 90 συστάσεις που δέχθηκαν από την καθολική περιοδική εξέταση του ΟΗΕ. Δεν είναι βέβαια δηλαδή οι πιο σημαντικές συστάσεις, γιατί είναι κυρίως συστάσεις που αφορούν τα παιδιά, τις γυναίκες και τους αναπήρους. Οι πιο σημαντικές βέβαια συστάσεις δεν έγιναν δεκτές από την κυβέρνηση της Ερυθρέας, όπως το θέμα των πολιτικών κρατουμένων, οι συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές. Όπως είπα, ανησυχούμε τα μάλα γιατί κατάσταση της φυλακές και μας προβληματίζει η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρόλο που διαπιστώνουμε κάποια βήματα πρόοδου. Όπως σας είπα, ο περιορισμός της στρατιωτικής θητείας είναι πολύ σημαντικό βήμα και θα πρέπει να εφαρμοστεί η σχετική υπόσχεση. Γιατί αυτή η απεριόριστη στρατιωτική θητεία είναι στους λόγους μαζικής εξόδου των Ερυθρέων από τη χώρα. Άλλο πρόβλημα είναι η έλλειψη οικονομικών προοπτικών για τους νέους και γενικώ για τον πληθυσμό. Και αυτό εξωθεί στη μετανάστευση. Θεωρούμε ότι ε, αυτά που επιδιώκουμε με την αναπτυξιακή μας βοήθεια και τη Συμφωνία του Κοτονού είναι να στηρίξουμε το λαό της Ερυθρέας. Δεν είναι κονδύλια που τροφοδοτούν τον προϋπολογισμό της χώρας. Είναι κονδύλια που χρηματοδοτούν συγκεκριμένα προγράμματα. είτε γεωργικά, είτε θέματα επισητιστικής ασφάλειας. Πρόκειται για προγράμματα που ουσιαστικά ωφελούν τον τοπικό πληθυσμό. Η συνάδελφος μπορεί να σας ενημερώσει πώς η αναπτυξιακή μας βοήθεια βοηθά το λαό της Ερυθρέας και δεν στηρίζει την κυβέρνηση της χώρας. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τη Συμφωνία του Κοτονού για να συνεχίσουμε τον πολιτικό μας διάλογο. Και είναι σημαντικό να συνεχιστεί ο διάλογος αυτός με την Ερυθρέα Ακριβώς επειδή ανησυχούμε ιδιαίτερως και για τη δυναμική που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί η Ερυθρέα έχει 1200 χιλιόμετρα ακτογραμμής στην Ερυθρά θάλασσα. Θα πρέπει να σταθεροποιηθεί η περιοχή. Υπάρχει το θέμα της Ιεμένης, του, της διαφοράς ε, των συνόρων ε, μεταξύ Ερυθρέας και Αιθιοπίας ε, δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα σύνορα. Επίση, ε, το πρόβλημα με το Νότιο Σουδάν. Θα πρέπει να υπάρξει μια σταθεροποίηση τη περιοχή. Γι' αυτό συνεχίζουμε την αναπτυξιακή μα συνεργασία με την Ερυθρέα και γι' αυτό θέλουμε και συνέχιση του διαλόγου με την Ερυθρέα. Στα τέλη Ιανουαρίου, ο ειδικό εκπρόσωπο ε, για το κέρα τη Αφρική ο κύριος Αλεξάνδρ Χόντος επισκέφθηκε την Ερυθρέα και είχε δύο ώρες συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας. Ε, συζητήθηκαν εκεί και περιφερειακά θέματα αλλά και εσωτερικά ζητήματα της Ερυθρέας. Οπότε εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι σημαντική η συνέχιση του διαλόγου και απαραίτητη και με την αναπτυξιακή μας ε, ε, βοήθεια προσπαθούμε να θέσουμε και το ζήτημα της οικονομικής διακυβέρνησης και ζητούμε μεταρρυθμίσεις από τη χώρα, γιατί η κυβέρνηση θέλει να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, αλλά με την ισχύουσα νομοθεσία είναι αδύνατο να το καταφέρει, γιατί είναι δύσκολο να ανοίξει κανείς επιχείρηση στην Ερυθρέα. Και οι περισσότεροι κλάδοι είναι κρατικοί. Ανήκουν στο κυβερνόν κόμμα και είναι δύσκολο να αναπτυχθεί ο ιδιωτικό κλάδο, οι ιδιωτικέ επιχειρήσει. Και για τι γυναίκε είναι δύσκολη κατάσταση. Οπότε και στο διάλογό μα θα θέσουμε και θέτουμε συνεχώ το ζήτημα τη οικονομική διακυβέρνηση, ευελπιστώντα ότι θα γίνουν και νομοθετικέ αλλαγέ και μεταρρυθμίσει. Τέλο, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, Πιστεύουμε ότι τα αίτια της μετανάστευσης ε, είναι καταρχήν η έλλειψη, η συρρήκνωση του πολιτικού χώρου και η πολύ δινή οικονομική κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του χαρτού, η Ερυθρέα ήταν ανέκαθεν υπέρ και ενδιαφερόταν ε, για τη διαδικασία του χαρτού γιατί η μαζική έξοδος ε, από τη χώρα προβληματίζει τις αρχές. Συμμετείχα ε, με ενεργά στην σύνταξη της ε, διακήρυξης για τη μετανάστευση στα πλαίσια της διαδικασίας του Χαρτούμ. Υιοθετήθηκε η διακήρυξη αυτή στα τέλη του Νοεμβρίου και προέβλεπε και στη σύσταση μιας ε, διευθυντικής επιτροπής. Η Ερυθρέα συμμετέχει σε αυτή την ε, επιτροπή και μαζί με το Σουδάν, τον Νότιο Σουδάν, την Τινησία συμμετέχουν στην επιτροπή. Αυτή από ευρωπαϊκής πλευράς ε, εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Αφρικανική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Επιτροπή αυτή θα αναπτυχθούν κάποιες μεθοδολογίες εργασίας, θα προσδιοριστούν κάποια προγράμματα προτεραιότητες και κάποιες πολιτικές προτεραιότητες. Μία από τις προτεραιότητες θα ήταν η εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους μετανάστες. Και ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων των μεταναστών με ε, ιδιαίτερη έμφαση τους ευάλωτους μετανάστες, τις γυναίκες και τα παιδιά. Η πρώτη συνεδρία αυτής της ε, Ειδική Επιτροπής ε, θα λάβει χώρα στα τέλη Απριλίου. Ξέχασα και την Αίγυπτο που επίσης είναι δραστήριο μέλος αυτής της ε, Διευθυντικής Επιτροπής. Αρχίζουμε με αργούς ρυθμούς, αλλά σταθερά αυτή τη διαδικασία. Ήδη μάλιστα έχουμε προβλέψει κονδύλια για το πρόγραμμα αυτό και τη λειτουργία αυτής της Επιτροπής και θα σας κρατούμε ενήμερους ε, για την πρόοδο και τα βήματα που θα γίνουν τους επόμενους μήνες. Αναφέρθηκε και μία ερώτηση για το κατά πόσο η κυβέρνηση Ερυθρέας στηρίζει και χρηματοδοτεί τρομοκρατικές ομάδες στη Σομαλία. Στην τελευταία έκθεση της ε, ομάδας παρακολούθησης Σομαλίας Ερυθρέας αναφερόταν για το θέμα αυτό ότι φαίνεται πως η κυβέρνηση έπαψε να στηρίζει τρομοκρατικές ομάδες ε, στη Σομαλία. Ή τουλάχιστον στην έκθεση αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, αποδείξεις που να τεκμηριώνουν τέτοιο ισχυρισμό. Βέβαια υπάρχουν και αντίθετες ε, απόψεις, κυρίως από την Αιθιοπία, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να στηριχθούμε στο περιεχόμενο της έκθεσης της ομάδας παρακολούθησης. Τουλάχιστον αυτά έλεγε η περσινή έκθεση. θα υποβληθεί και φετινή έκθεση. Θα δούμε τα πορίσματά της, γιατί η Αιθιοπία αφισβήτησε τα πορίσματα της προηγούμενης έκθεσης. Θα δούμε την επόμενη, ίσως φέτος, ε, οι μυστικές υπηρεσίες της Αιθιοπίας βοηθήσουν. Πάντως είναι δύσκολο να αποδειχθεί στήριξη, χρηματοδότηση τέτοιων τρομοκρατικών ομάδων. Πάντως η Επιτροπή Παρακολούθηση απεφάνθη ότι δεν έχει στοιχεία που να τεκμηρώνει τέτοιο ισχυρισμό. Εμείς ευχαριστούμε. Ακούσουμε και από την ΤΕΦΚΟ και επίση ε, σύμφωνα με όσα μα είπατε να δούμε τι έχουν να σχολιάσουν προσκεκλημένοι μα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΤΕΦΚΟ. Ευχαριστώ όσον αφορά τώρα την συνεργασία. Χωρί να μακρηγόρω να σα πω τι έχει γίνει. Πρόκειται για τα προγράμματα του 10ου ΦΕΔ, το 10ο ΦΕΔ, το οποίο ε, στην αρχή είχε προκοδότηση 120 εκατομμύριων ευρώ, αλλά κατόπιν έγινε περικοπή και κατέβηκε στα 52 ε, ευρώ. Οπότε δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη περικοπή του αρχικού ποσού που είχε διατεθεί. Τώρα όσον αφορά ε, αυτό το ποσό, 40 εκατομμύρια αφορούν την γεωργία για να βελτιωθούν τα ζητήματα άρδευσης και τις μερικές περιοχές να μπορούν να μονοκαλλιεργήσουν, να υπάρχει διατροφική ασφάλεια γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα τέτοιο στην ε, Ερυθρέα. Όμως, μια που δεν ήταν ελεύθερη πρόσβαση στη χώρα, δεν μπορέσαμε να αξιολογήσουμε ακριβώς τη διάσταση του προβλήματος. Όμως, σαφώς υπάρχει το πρόβλημα. το πρόγραμμα αυτό σιγά σιγά άρχισε να τρέχει, είπαμε 40 εκατομμύρια, πάρα πολύ λίγα λεφτά έχουν εκταμιευθεί από τότε και ανεστάλλει η συνεργασία από την κυβέρνηση μονομερός το 2011 και τώρα τρέχει το πρόγραμμα για βοήθεια προς την κυβέρνηση της χώρας, για την διοίκηση, αλλά εκεί υπάρχουν προβλήματα. Γιατί Ακριβώς τώρα υπάρχει ε, διαρροή εγκεφάλων από τη χώρα. Δηλαδή φεύγουν από τη χώρα εκείνοι οι οποίοι ήταν οι πτυχιούχοι. Πρόβλημα συνεργασίας μόνος υπάρχει, αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα ε, το, όσον αφορά τα τοπικά δικαστήρια, community courts. Να δούμε πώς σε τοπικό επίπεδο μπορούμε να στηρίξουμε τη δικαιοσύνη, γιατί βέβαια θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τι γίνεται με τα προγράμματα, βεβαίω με τα προγράμματα να μην κάνουμε κάτι αντίθετο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ούτε να χρησιμοποιούμε τα προγράμματα αυτά από το κράτο με τρόπο που δεν θέλουμε. Αλλά αυτό πάλι είναι δύσκολο να το διαπιστώσουμε. Μια, ένα μικρό άνοιγμα έγινε όσον αφορά κάποια πολύ μικρά προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να υποστηρίξουμε κάποιε σχετικέ πρωτοβουλίε. να βοηθήσουμε κάποιους ε, φορείς αθλητικούς, ε, φορείς για τις γυναίκες, φορείς ε, αναπήρων και δεν πρόκειται για κυβερνητικούς φορείς, πρόκειται για κάποιους νόσους προσώπων που δρούν σε τοπικό επίπεδο. Οπότε να δημιουργηθεί μια απαρχή κοινωνίας πολιτών με αυτόν τον τρόπο. Κάτι άλλο τώρα που αφορά τον διάλογο με σκοπό την συνεργασία τονίζουμε την έλλειψη αποτελεσμάτων, γιατί χρειάζεται η Ερυθρία να κάνει ένα άνοιγμα, να κάτι να γίνει με τους πολιτικούς κρατουμένους. Αν δεν γίνει κάτι με τους στόχους της χιλιετίας και να γίνει άνοιγμα προς την αξιολόγηση στη χώρα. Και κάτι άλλο τώρα που προσπαθούμε ε, να τους πούμε είναι μια προσπάθεια συνεργασίας με τις γείτονες χώρες, να υπάρξει περισσότερη περιφερειακή ολοκλήρωση, να βγει η χώρα από την πολιτική απομόνωση, να δοθούν οικονομικά κίνητρα, οπότε αυτό ίσως θα μπορούσε να αλλάξει προς το καλύτερο την κατάσταση της χώρας. Άρα αυτό θέλουμε. Γι' αυτό και συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης για να υπάρξει αυτός ο διάλογος για τη συνεργασία και έτσι να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις για την πολιτική κατάσταση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εν γέννη. Όμως, είπαμε, η πρόοδος είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Αλλά δεν υπάρχουν ούτε αυτές οι μικρές σταγόνες συνεργασίας, ε, τότε δεν μπορούμε να έχουμε κανένα είδους διάλογο ή πρόσβαση στη χώρα. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Αν θέλετε ένα σύντομο σχόλιο γι' αυτά, παρακαλώ, κυρία Κίτερουτ. Ευχαριστώ. Θέλω πολύ σύντομα να πω ότι με χαρά ακούω ότι περιορίστηκε στους 18 ε, μήνες η εθνική στρατιωτική θητεία. Τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει να περάσουν 18 μήνες όμως για να βεβαιωθούμε ότι αυτοί που επιστρατεύτηκαν τώρα θα απολυθούν. Ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα. Εδώ έχουμε να κάνουμε πολύ σημαντικά θέματα. Αν δούμε λοιπόν τελευταία έκθεση από το Συμβούλιο, βλέπουμε ότι η θητεία ισοδυναμεί με αναγκαστική δουλεία. Θέλω λοιπόν να δω να υλοποιείται αυτή η αλλαγή με συγκεκριμένα βήματα. Για τους λίγους δημοσιογράφου που έχουν ε, αποφυλακιστεί. Χαίρομαι. Πολύ. Πολύ καλά νέα. Αλλά πώς σημαίνουν ακόμα στη φυλακή. και πολλά άλλα πράγματα θα είχα να αναφέρω. Θα επικεντρωθώ όμως σε κάτι άλλο. Τα κοινοτικά δικαστήρια, πολύ καλή ιδέα να έρχονται κοντά στους ανθρώπους, κοντά στους πολίτες, αλλά που βρίσκονται οι νόμοι πάνω στους οποίους στηρίζονται για τη λειτουργία τους και πώς εξασφαλίζεται η ορθή διεξαγωγή της δίκης. Και κάτι το οποίο δεν έθιξα είναι όμως πολύ σημαντικό πιστεύω σε όλη αυτή τη συζήτηση για τους νέους που εγκαταλείπουν τη χώρα. Υπάρχει γνήσια ανάγκη για προσφορά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά τη θητεία. Και το λέω με ποια έννοια. Ότι ο νέος 17-18 όταν πάει στη λεγομενη δωδεκάτη τάξη όπως ονομάζεται, τι συμβαίνει, χρειάζεται τρεις μήνες στρατιωτική εκπαίδευση στο στρατόπεδο πριν περάσει τις τελικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι συνδεδεμένο απόλυτα το να κάνει αυτό το τρίμηνο της εκπαίδευσης. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι πολλοί οι νέοι που δεν μπορούν να τελειώσουν και να προχωρήσουν σε τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Αυτοί που φτάνουν λοιπόν στο τέλος της ε, ε, δευτεροβάθμιας και πρέπει να κάνουν το τρίμηνο, πολλές φορές επιλέγουν στο τέλος τη στρατιωτική εκπαίδευση και τη στρατιωτική σταδιοδρομία. Αυτό, αυτή την διασύνδεση πρέπει να την ε, κοιτάξουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Και πρέπει για να ολοκληρώσω να πω ότι χρειάζεται να, δούμε ότι οι Ερυθρέοι αισθάνονται ασφαλείς στην ίδια τους τη χώρα, να μην κινδυνεύουν από αυθαίρετη κράτηση, φυλάκιση, ε, χωρίς δίκαιη δίκη η οικία τους. Χρειάζεται να ανοικοδομηθεί αυτή η εμπιστοσύνη από το λαό. Η εμπιστοσύνη που θα αισθάνεται ο λαός για την κυβέρνησή του και πρέπει να το κάνει αυτό η κυβέρνηση αυτό. Και βέβαια υπάρχουν και πολλά πρέπει να κάνει η διεθνής κοινότητα για να βοηθήσει. Αυτό όμως ε, είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Εκεί εντοπίζονται τα προβλήματα και σταματάω εδώ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Σύντομο σχόλιο για την θητεία. Δεν έχω δει πουθενά επίσημη δήλωση από την κυβέρνηση που να δηλώνει ότι θα τηρήσει τις ε, ε, διατάξεις που αφορούν την θητεία. Το μόνο που έχουμε ως δεδομένο είναι ότι κάποιος δήλωσε από τη Βρετανία ότι ένας ανώτερος αξιωματούχος του είπε «Σε αυτό θα στηριχθούμε». Έχουμε ανθρώπους που βρίσκονται επιστρατευμένοι από το 1994. Γιατί δεν αρχίζουν να αποστρατεύονται, γιατί δεν ε, τους απολύουν. Γιατί να περάσουν άλλου 18 μήνε. Αυτό, είναι πάρα, Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν μιλώ για ανάπτυξη των, ε, και επανάληψη των σχέσεων και των συνομιλιών. Πολύ σημαντικό. Αλλά η μέθοδος του ραβδιού και του κινήτρου, του, του κινήτρου και της κυρώσεως είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορούν να χρησιμοποιούν λοιπόν την θητεία για πρόσχημα και να την αξιοποιούν σε μία παγωμένη σύγκρουση με την Αιθιοπία. Πρέπει η εθνική κοινότητα να εμπλακεί στην υπόθεση αυτή. Πρέπει να αναπτυχθεί μια ουδέτερη επιτροπή συνόρων που ήδη έχουν συμφωνήσει δύο χώρες και να αποσύρει η Αιθιοπία τα στρατεύματά της από τα σύνορα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, κυρώσεις. Οι κυρώσεις είναι ε, συμβολικές και ενδεικτικές των διπλών μέτρων και σταθμών που, χρησιμοποιούν που χρησιμοποιεί το Συμβούλιο. Δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι αντιπαραγωγικά ή τι άλλο. Πρόσβαση στα όπλα. Ε, όποιος έχει λεφτά μπορεί να βρει όπλα, ό,τι θέλει, στη μαύρη αγορά. Είναι γνωστό αυτό. Άρα χρειάζονται ένα-δυο κίνητρα για να, προσ... για να προσεγγίσετε το καθεστώς μέσα από τις συνομιλίες να πούμε αποστρατιωτικοποιήστε την εκπαίδευση. Αντί να κλείνουν όλα τα πανεπιστήμια γιατί κάποιος συνέκρινε την ε, Ερυθρέα με τη Βόρεια Κορέα. Όχι. Η Βόρεια Κορέα είναι πολύ καλύτερη. Θα φέρω αντι... αντιρρήσεις εδώ. Η Βόρεια Κορέα παράγει πυρηνικούς επιστήμονες. Εδώ έχουν κλείσει το μόνο πανεπιστήμιο της χώρας και το έχουν αντικαταστήσει από ένα συνονθήλευμα ε, σχολών, οι οποίες δεν φτάνουν το επίπεδο της δευτεροβάθμιας. Ήταν λοιπόν κάπως ε, προχωρημένη αυτή η σύγκριση. Λοιπόν, με κίνητρα και με κυρώσεις, έναντι του καθεστώτος, μπορούν να φύγουν τα ζητήματα και να τεθούν θέματα πολιτικού διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, περιεκτική και θέλουμε να υπάρξει και συνέχεια. Αργότερα στο διευρυμένο Προεδρείο θα πρέπει να δούμε δεδομένης και τις επικείμενης συμφωνίας του Κοτονού ε, την ε, πιθανότητα να συντάξουμε ψήφισμα. Για το τελευταίο μας ψήφισμα για το θέμα αυτό ανάγεται στο 2011. Να δούμε λοιπόν αν είναι σκόπιμο να συντάξουμε νέο ψήφισμα. Εν πάση περιπτώσει με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά που ήρθατε. Έχει καταθέσει το μεταξύ και ο ειδικό ηγητή ε, των Ηνωμένων Εθνών για του ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. τόσο λίγο θα περάσουμε στο δικό του θέμα.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 Λοιπόν, συνεχίζουμε. Περνάμε στην ανταλλαγή απόψεων με τον Μισελ Φόρς, τον ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τους ακτιβιστές συγκεκριμένα ανθρώπινα δικαιώματα. με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στη συνεδρίασή μας τον Μισελ Φόρστ, ε, τον ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων ε, για τις ε, συνθήκες το, της άσκησης των δραστηριοτήτων της υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα θέμα που συχνά απασχολεί την Επιτροπή μας και μάλιστα πέρυσι είχαμε την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο ε, εγκρίθηκε στο Στρασβούργο και μία από τις συστάσεις ε, της έκθεσης αυτής προέβλεπε και τις κατευθυντήριες γραμμές, ε, προέβλεπε την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να εφαρμοστούν. Επίσης, ζητήσαμε και προβλέψαμε σύσταση ειδική ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να είμαστε διαρκώς ενήμεροι για την κατάσταση και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Έχουμε και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, οπότε χρήσιμο θα ήταν να έχουμε και εσείς και εμείς άμεση ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Φόρστ. Ευτυχώς έχουμε αρκετό χρόνο, οπότε θα προλάβουμε, πιστεύω, να Υποβάλλουμε και εμείς, αλλά να δώσουμε την ευκαιρία και σε εσά ε, να θέσετε απευθείας ερωτήματα στον κύριο, στον κύριο Φόρστ, ο οποίος ανέλαβε πέρυσι τα καθήκοντά του. Μάλιστα είχαμε προηγουμένως ε, συνάντηση με την προκάτοχό σας, την κυρία Μάργαρετ Σεκαγκάια. Ε, είναι πολύ καλή αυτή η παράδοση που έχει δημιουργηθεί στην Επιτροπή μας για συνεργασία με τον ειδικό εκπρόσωπο, ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χάρη στη συζήτηση που θα έχουμε θα ενημερωθούμε για τις προτεραιότητές σας ε, στη νέα σας θητεία, αλλά θα πρέπει να δούμε και τη στρατηγική μας και τις πολιτικές μας ε, για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα αύριο θα έχετε ανταλλαγή απόψεων ε, με την ΚΟΧΟΜ, την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολύ συχνά έχουμε συναντήσει με εκπροσώπους της ομάδας αυτής για να συντονίζουμε τις πολιτικές μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε θα ξεκινήσουμε με τη δική σας παρουσίαση, θα ακολουθήσει συζήτηση. Έχουμε και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύο μάλιστα, Διγκίση και Νορμό. Θα ακούσουμε και τη δική τους παρέμβαση και έχουμε και εκπρόσωπο της ΑΕΔ, τον κύριο Γκάρντ Μπράιαν, αν δεν κάνω λάθος. Και φυσικά μετά οι βουλευτέ θα υποβάλλουν ερωτήσει. Κύριε Φόρστ, είπατε θα μιλήσετε γαλλικά, δεν κάνω λάθο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, όντω. Θα μιλήσω γαλλικά, γιατί αυτό μου σύστησε η κυβέρνηση. Να χρησιμοποιώ τη γαλλική στι διεθνεί διασκέψει, ώστε να παραμείνω τα γαλλικά μία από τι ε, πρωταρχικές γλώσσε εργασίας και των Ηνωμένων Εθνών. Πρόεδρε, κύριοι πρέσβοι, εξοχότατοι, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτέ. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που μου δίνετε μερικά λεπτά για να σας παρουσιάσω το περιεχόμενο των πρώτων ερευνών και εργασιών μου μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου και να έχουμε και ανταλλαγή απόψεων και διάλογο γιατί θα χρειαστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως ε, έχουμε ανάγκη και τα Εθνικά Κοινοβούλια και αν μου επιτρέπετε θα υποβάλω κάποιες συστάσεις ε, στην παρουσίασή μου για την καλύτερη στήριξη που μπορούμε να έχουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χάρη στη βοήθεια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Γενικής Διεύθυνσης ΤΕΦΚΟ και ευχαριστώ επ' ευκαιρία τον Πατρίς Λεωνορμό, πριν μερικούς μήνες ξεκινήσαμε μια σειρά περιφερειακών διαβουλεύσεων. Όταν ανέλαβα πέρυσι τον Ιούνιο το καθήκοντά μου, οι διεθνείς οργανώσεις ε, μου ζήτησαν πρώτα απ' όλα να ακούσω τις ανάγκες των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και χάρη στον προπολογισμό της ΔΕΦΚΟ είχα 7 περιφερειακές διαφουλεύσεις με ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την περιοχή του Περσικού Κόλπου, από την Βόρεια Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη, Κεντρική Αφρική, Λατινική Αμερική και μου έχουν απομείνει δύο ακόμη περιφερειακές διαβουλεύσεις μία στην Ανατολική και μία στη Δυτική Αφρική. Και πιστεύω ότι χρήσιμο θα ήταν να γίνει μια διαβούλευση και με ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Δυτικής Ευρώπης, ε, ε, του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Γιατί και στις χώρες μας ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες οι ακτιβιστές πολλές φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα με κανόνες και νομοθετικές διατάξεις που ποινικοποιούν τη δραστηριότητά τους. Χάρη σε αυτές τις περιφερειακές διαβουλεύσεις θα κάνω μια ανάλυση των εθνικών και των περιφερειακών τάσεων, θα κάνω μια εκτίμηση των απειλών κατά ειδικών ομάδων και θα, και θα αξιολογήσω την αποτελεσματικότητα εθνικών και περιφερειακών μέτρων για να εξασφαλίσουμε καλύτερη προστασία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίση, ε, ε, ελπίζω τα επόμενα χρόνια να απτυχθούν νέε μέθοδοι προστασία των ακτιβιστών. Αυτά θα είναι το αντικείμενο και τη επόμενη μου έκθεση ε, που θα υποβάλω τον επόμενο Οκτώβριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και μετά από επιτόπιες διαβουλεύσεις, μετά από ακροάσεις των ακτιβιστών θα υποβάλω τις συστάσεις μου στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ για την κατάσταση προστασίας των ακτιβιστών και τις ανάγκες για το μέλλον, γιατί η μέχρι τώρα κατάσταση δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ακτιβιστών. Μέχρι στιγμή ε, συνάντησα πάνω από 350 ακτιβιστές ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων από 70 διαφορετικές χώρες, αποφασισμένους ε, και θαραλέου άνδρες και γυναίκες που μου περιέγραψαν τις απειλέ τις επιθέσεις, τους φόβους, τις προσδοκίες τους από την θητεία μου, από τους ίδιου, αλλά και από τη διεθνή κοινότητα ηγένη. Όλοι αυτοί οι ακτιβιστέ που συνάντησα στι περιφερειακές διαβουλεύσεις και που καθημερινά μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε πόσες απειλές δέχονται, εκφοβισμούς, βρίσκονται στο στόχαστρο επιθέσεων, γίνονται θύματα παρενόχλησης, ποινικοποίηση, θύματα συκοφαντικής δυσφήμισης και δεν μπορούν να εκφράσουν την γνώμη τους ελεύθερα ή να συναθρίζονται ελεύθερα. Και παρόλα αυτά συνεχίζουν τις ε, ε, θαραλές ε, δραστηριότητες προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μερικοί βέβαια δυστυχώς ε, συλλαμβάνονται, κρατούνται, βασανίζονται, ξαφανίζονται, αγνοείται η τύχη τους οι παραβιάσει είναι διαφορετικές με τι διαφορετικές χώρες ή περιφέρειες, αλλά στόχο του είναι να απαξιώσουν, να φημώσουν και να εξοντώσουν σε τελική ανάλυση του ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ θα επικεντρωθώ σε ορισμένα σημεία που χρήσουν προσοχή κατά τη γνώμη μου, γιατί όπω σα είπα, του επόμενου μήνε και χρόνια θα χρειαστώ τη δική σα υποστήριξη θα χρειαστώ πραγματικά και τη βοήθεια των Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και των Περιφερειακών Κοινοβουλίων. Από τις πρώτες συναντήσεις που είχα με ακτιβιστές στη Γενέβη τον περασμένο Ιούνιο, ανέκυψε η προφανής ανάγκη να επικεντρώσω τη θητεία μου στην προστασία των, των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι οι πιο εκτεθειμένοι και αντιμετωπίζουν τις περισσότερες απειλές και κινδύνους. Είναι κυρίως οι ακτιβιστές που προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών και προσπίζουν τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των ακτιβιστών ε, ΛΟΑΔΜ, των ακτιβιστών Προστασία ταυτότητα του φύλου, γιατί αυτές, αυτοί οι ακτιβιστέ ε, απειλούνται ιδιαίτερα. επίση και τους οικολόγους ακτιβιστέ, που ασχολούνται με τα δικαιώματα του, ε, των ανθρώπων σε επιχειρήσει, αλλά και αυτών που καταγγέλουν συγκεκριμένε παραβιάσεις, η κρού τον κόδωνα του κινδύνου. Μερικέ φορέ δεν έχουν καν το δικαίωμα ελεύθερη συνάθρηση ε, οι ακτιβιστέ. Υπάρχουν περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό που είναι αδικαιολόγητοι. Γι' αυτό και όλο και περισσότερο έχω στενή συνεργασία με του άλλου ειδικού ε, εισηγητέ ε, που ασχολούνται με το δικαίωμα έκφραση, ελευθερίας έκφρασης και ελευθερία συνάθρηση. Πιστεύω ότι καλύτερα να έχουμε συνεργασία μεταξύ μα, αντί ο καθένα να δρά απομονωμένα. Χρειάζεται συντονισμό για να υπεθυμίζουμε το διεθνέ δίκαιο και την ανάγκη ε, συνεχούς προστασίας των ακτιβιστών. Επίσης ε, θα συνεργαστώ και με τους ε, άλλους ειδικού συγητές των περιφερειακών οργανώσεων, της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Αφρικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών. Και πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε στο Παρίσι μία συνάντηση στην οποία προσκάλεσα και τον Ήρσμι Μινίκα, τον ειδικό επίτροπο του Συμβουλίου τη Ευρώπης και τον κύριο Λαμπρινίδη για να δούμε από κοινού τι δυνατότητες έχουμε για κοινή δράση σε ευαίσθητα θέματα ή σε πιο ε, ανησυχητικά ε, για τους ακτιβιστές ε, ζητήματα για να έχουμε μια κοινή προσπάθεια. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε κοινή δράση για να καταπολεμήσουμε την αντιμορρησία που είναι από τις βασικότερες μάστιγες των ακτιβιστών. Επίσης, είχα συναντήσεις και με άλλους ενδιαφερομένους προκειμένου να ξεκινήσουμε νέες δράσεις για να ενισχύσουμε την εφαρμογή της οικομενικής Διακήρυξης του ΟΗΕ για τους ακτιβιστές αλλά και τις κατευθυντήρες γραμμές του ΟΗΕ για τους ακτιβιστές. Επίσης, τις κατευθυντήρες γραμμές του, της ΟΑΣΕ ε, γιατί όλο και περισσότερες χώρες ε, εκπονούν τις δικές τους κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των ακτιβιστών. Πάντως πιστεύω ακράδαντα στην συνεχή συνεργασία και τον επικοδομητικό διάλογο με τις κυβερνήσεις ε, ε, και τις επιμέρους χώρες. Γιατί η θητεία μου θα έχει μόνο στόχο την καταγγελία και τη στυλίτευση, αλλά και την πρόταση απτής συνεργασίας με τις διάφορες χώρες που θα στηρίξουν αυτή την εντολή. Γι' αυτό και θα προτείνω την έναρξη πολλών πρωτοβουλειών. Τώρα, με απασχολεί ιδιαίτερο το μικρό ποσοστό εφαρμογής των συστάσεων των διαφόρων φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΙΕ και των μηχανισμών που υπάρχουν για την προστασία των ακτιβιστών σε διεθνές επίπεδο. Θα μιλήσουμε αργότερα για τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό. Θα μιλήσω και το απόγευμα στη συνάντηση που θα έχουμε την ΤΕΦΚΟ και αύριο στη συνάντηση με την ομάδα εργασία του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά, την ΚΟΟΜ. Πιστεύω ότι δεν, θα δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε στρατηγικέ και μηχανισμού για να προστατεύσουμε καλύτερα του ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν δεν ενισχύσουμε την εφαρμογή των μέτρων. Θα προσπαθήσω να πείσω τι κυβερνήσει ε, να εφαρμόσουν ε, τα καλύτερα παραδείγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τα λάβουν υπόψη στις εθνικές νομοθεσίες, ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα, ε, για να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή των συστάσεων των δύο προκατόχων μου, των δύο προηγούμενων ειδικών εισηγητών, ε, θα πραγματοποιήσω σύντομες επισκέψεις ε, παρακολούθησης ε, σε χώρες που είχαν επισκεφτεί και οι προκατοχή μου για να δω κατά πόσο εφαρμόστηκαν οι προηγούμενες ειδικέ του συστάσεις και να καλέσω τις, την κοινωνία των πολιτών, τους εθνικούς φορείς και τις εθνικές οργανώσεις να εφαρμόσουν τις συστάσεις των δύο προηγούμενων ειδικών εισηγητών. Θα έχω σύντομες επισκέψεις σε διάφορες χώρες και θα δεχτώ και προσκλήσεις πολλών χωρών Εκεί θα έχω συνάντηση με πανεπιστημιακούς, θα λάβω μέρος και σε πάνελ συζήτησης με ακτιβιστές και όλα αυτά με απόλυτο σεβασμό των κανόνων του κώδικα διοντολογίας που διέπει τη θητεία μου και φυσικά θα ενημερώνω τη Γενέβη για τις διάφορες συναντήσεις που θα έχω. Επίσης θα βλέπετε στην έκθεσή μου ανακοινωθέντα με όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις ε, που έλαβα από τις χώρες. Θέλω διαφάνεια για να μπορούμε να παρακολουθούμε και τις μεμονωμένες υποθέσεις και τις ε, καταστάσεις αναχώρα. Έχουμε εκθέσεις αναπεριφέρεια αλλά και αναχώρα με ανάλυση των περιφερειακών τάσεων και των κρατικών τάσεων. Με τις ανακοινώσεις αυτές θα παρακολουθούμε το βαθμό συνεργασίας των διαφορών χωρών με τα διάφορα φόρα των Ηνωμένων Εθνών. Πέρυσι δώσαμε σε 84 χώρες 231 συστάσεις ε, για 530 ακτιβιστές, 119 από αυτούς ήταν γυναίκες ακτιβίστριες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έλαβα 128 απαντήσεις από τις χώρες, δηλαδή 55% ποσοστό απαντήσεων, αύξηση μικρή σε σχέση με πέρυσι. Αυτό που ανησυχεί είναι ότι στις ανακοινώσεις αυτές 28 ε, αφορούσαν ε, σχέδια, ε, σχέδια εθνικά που κατά τη γνώμη μου ε, θα ασκήσουν αρνητικό αντίκτυπο και θα επηρεάσουν αρνητικά το περιβάλλον εργασίας και τις συνθήκες δραστηριότητας των ακτιβιστών. Είχα φυσικά στενή συνεργασία με τους ε, δύο συναδέλφους ε, ειδικούς ηγητές, κ. Μανεκάη, ε, την ειδική συγγήτρια για την ελευθερία του συνα... της συνάθρησης και ίσως και σε αυτό το θέμα θα μπορούσε να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δούμε με ποιο τρόπο και τα εθνικά κοινοβούλια θα υποβάλουν νομοθεσίες που δεν θα εμποδίζουν όπως έχει γίνει μέχρι τώρα το έργο των ακτιβιστών. Έστειλα και αυτό είναι ακόμη πιο ανησυχητικό, 32 ανακοινώσεις ε, για αντίπεινα που έχουν εφαρμοστεί εις βάρος ε, ε, ιδιωτών ή ομάδων εξαιτή συνεργασίας τους με τα κράτη-μέλη. Αυτές οι ανακοινώσεις αφορούσαν ακτιβιστές που ήταν θύματα ε, συκοφαντικής δυσφήμισης, απαγόρευσης μετατόπισης, εκφοβισμού, παρενόχλησης, ε, ψυχοφαντικής δυσφήμισης, άρνησης ε, ε, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ε, καταχρηστικής αυθαίρετης κράτησης, άμεσων απειλών, φυσικών, σωματικών επιθέσεων και μερικές φορές ακόμη και δολοφονιών. Αυτές οι ανακοινώσεις τράφηκαν σε προς 22 χώρες, τις οποίες θα παριθμίσω, γιατί σε αυτές θα πρέπει να επικεντρωθείτε για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στη Σαουδική Αραβία και στον Παχρέν, στην Κίνα, ε, στην Κούβα, στην Αίγυπτο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στην Ρωσική Ομοσπονδία, στην Ονδούρα, την Ινδία, το Ιράν, τη Μαλαισία, Μαλδίδες, Μεξικό, Μιανμάρ, Ομάν, Πακιστάν, Σρι Λάγκα, Συρία, Τατζικιστάν, Ταϊλάνδη, αλλά και στο Βιετνάμ. Και αυτό το είπαμε δημοσία φέτο, ενώπιον τη Γενική Σύλληψη του ΟΗΕ και την περσμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και θέλω να το επαναλάβω εδώ, ενώπιον ημών επισήμω και αποφασιστικά ότι πρόκειται για κάποιε πράξει αφόρητε, απαράδεκτε, για τι οποίε είμαι πάρα πολύ προβληματισμένο και ανησυχώ, γιατί έχουμε όλο ένα και περισσότερο τέτοιε πράξει ε, εκφοβισμού ε, και αντιπίνων ε, κατά των όσων παλιών τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, άρα θα πρέπει κάτι να γίνει από τον ΟΗΕ ή και με τις ε, περιφερειακές οργανώσεις. Μιλούμε για αυτές τις εκστατείες συκοφάντησης, για άμεσων απειλών, σωματικών επιθέσεων, ανθρωποκτονιών και όλα αυτά ακόμα πιο συγκλονιστικά και εντυπωσιακά όταν προέρχονται από κάποιο χώρο που μετέχει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και έγινε αυτό με το Βιετνάμ και ο συγκεκριτής για τα θέματα συνείδησης και υγείας συνελήφθη όταν πήγε στο Βιετνάμ και η κοινωνία τον εμπόδισε να μπορέσει ε, να συναντήσει ε, όποιον ήθελε και οπότε και είχαμε επεισόδιο στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιωμάτων. Οπότε είχαμε αυτή την ε, κατέληξε το Συμβούλιο ότι δεν είναι δυνατόν τα κράτη να παροχλεί αυτούς που συμμετέχουν σε εργασίες του Συμβουλίου γιατί πρόκειται για κάποιες απειλές οι οποίες εξαπολύνονται κατά αυτών των αγωνιστών οπότε παρακαλώ και εσείς να διαβιβάσετε στα κράτη σας αυτό το μήνυμα στις κυβερνήσεις ούτω ώστε στο Συμβούλιο δικαιωμάτων να μην ανέχονται τέτοια αντίπεινα κατά των όσων αγωνίζονται για ανθρώπινα δικαιώματα ο οι ε, διεθνείς κοινότητες εξαρτώνται 100% από την ε, συνεργασία, τη συνεργασία την ανεμπόδιστη με την κοινωνία των πολιτών. Χωρίς μια τέτοια συνεργασία το έργο αυτών των οργανισμών και του ΟΗΕ δεν θα έχει ε, νοημοποίηση. Επομένω, επιγόντω θα πρέπει να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτέ τι επιθέσει, εκφοβισμό των αντιπίνων. Και κατακλείδη, κύριε Πρόεδρε, Παρακαλώ οι ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν όσο μπορούν περισσότερο αυτό το ψήφισμα 24 24 που τώρα βρίσκεται προς συζήτηση στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με αυτό το ψήφισμα λέμε για τη συγκρότηση μηχανισμού στον ΟΗΕ, ούτως ώστε να προστατεύονται όσοι υπερασπίζονται τα δικαιώματα ε, και αυτό να γίνεται με κάποιο φορέα νοτό του παρά το γενικό γραμματεία, ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται αυτά τα αντίπεινα και αυτέ οι απειλέ. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθούμε τι κάνετε και τι σχεδιάζετε. Για να δούμε λίγο το χρόνο μας. Μπορούμε από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να δούμε ποιος ενδιαφέρεται να λάβει το λόγο. Ωραία. Θα τα καταφέρουμε φαντάζομαι. μη κυβερνητικέ οργανώσει. Ζήτησα μόνο γιατί μια και έχουμε τον ειδικό εισηγητή, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή ευκαιρία. Λουτσία Ντεγκίζη και Λενόγμα θα είναι οι επόμενοι ομιλητές. Θα μας μιλήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα κύριος Λενομό νομίζω εκπροσωπεί την Επιτροπή, δεν είναι. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Καταρχάς θα ευχαριστήσω τον εισηγητή για τα λόγια του. Είναι πολύ δύσκολη η εντολή ε, και πολύ φιλόδοξη, με πολύ περιορισμένα μέτρα. Μέσα. Η υπερασπίση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα μέσον και για, την, ε, για τον αγώνα μας θα συνεχίσουμε να τον υποστηρίζουμε και τους αγωνιστές αυτούς αλλά και τον ίδιο τον εισηγητή. Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να προσθέσω από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ότι υποστηρίζουμε περίφραστα τον ρόλο του ειδικού εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήμασταν πάντοτε υπέρ ε, τη της δουλειάς που κάνει από τη θέση αυτή. Έχουμε παρακολουθήσει και με την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις περιφερειακές διαπραγματεύσεις. Καλωσορίζουμε την ε, προσέγγιση και εν ώψη των κυρώσεων από τον ειδικό εισηγητή. Θέλουμε και εμείς να δουλέψουμε στην κατεύθυνση αυτή και θα ήθελα να προσθέσω ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για την βελτίωση των συνθήκων για τους αγωνιστές των δικαιωμάτων. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από το Συμβούλιο των, των Γενικών Υποθέσεων ε, με την επέτειο των κατευθυντηρίων γραμμών τον προηγούμενο Ιούνιο. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε ότι πρέπει να εστιαστούμε στις γυναίκες αγωνίστρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιφερειακές και από μονομένες κοινότητες, δηλαδή στις πιο ευάλωτες ομάδες και νομίζω ότι αυτό ακολουθεί και τις επιλογές του ειδικού εισηγητή και νομίζω ότι έτσι μπορούμε και μετά τις καθημερινές γραμμές να πούμε ότι έχουμε προχωρήσει ιδιαίτερα και έχουμε υποστηρίξει τις ε, κοινότητες των αγωνιστών όπου, όπου δι, ε, προβαίνουμε σε δηλώσεις. Έχουμε προαγάγει σημεία εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και επικοινωνία σε κάθε τρίτη χώρα. Πάντα βεβαίως υπάρχει δουλειά που μένει να γίνει. Και θα κοιτάξουμε να βελτιάσουμε ακόμη περισσότερο τη δουλειά μας με τους αγωνιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου επιμερισμού του φόρτου και του έργου και της καλύτερης επικοινωνίας με απομονωμένες ή περιφερειακές ε, ομάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπράιον. Ο κύριος Λενορμό, αν μου επιτρέπει να διατυπώσω μια ερώτηση. Ναι, και είπε Μισελ στην αρχή ότι είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό της υλοποίησης των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας απασχολεί αυτό. Εννοείται χαμηλό επίπεδο υλοποίηση των συστάσεων από σώματα και φορείς των Ηνωμένων Εθνών. Όχι, από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον εγώ από την Τερμηνία λέει πρόεδρος είναι των ευρωπαϊκών συστάσεων σε σχέση με τις χώρες αυτές. Ναι, αν μου επιτρέπετε να παρεμβώ. Υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα. Καταρχάς έχουμε να κάνουμε την υλοποίηση των συστάσεων το UPR των ειδικών εισηγητών το, από τα κράτη-μέλη. Αλλά υπάρχουν και ζητήματα που προκύπτουν κατά τις διαφουλεύσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές κατευθυντηρίες γραμμές μπορούν να υλοποιηθούν από τις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες στα κράτη-μέλη. Είναι και αυτό κάτι το οποίο θα ε, οφείλαμε να συζητήσουμε. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να σας ενημερώσω για την έκβαση αυτών των συζητήσεων και με την Επιτροπή των Συνταγματικών είχα να το συζητήσω αυτό για σήμερα το απόγευμα και μπορούμε να συνεχίσουμε και αύριο αν θέλετε. Ναι, ευχαρίστως να γίνει αυτή η συζήτηση και εμείς τη θέλουμε βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις ως προς την υλοποίηση των κατευθυντηριών γραμμών. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Κατά τα άλλα, αυτά είναι όλα ζητήματα τα οποία συζητούμε πάντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Κύριος Παντσιέρη έχει στήσει το λόγο. Παντσέρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ψήσω την προσοχή του κύριου Φόρστ, του καλεσμένου μας, σε κάποια θέματα, γιατί και εγώ συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ κομβικό το ζήτημα των όσων αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ άλλων Υπήρχε ένα σημαντικό κομμάτι στην ετήσια έκθεση εκείνη που εγκρίναμε την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επρόκειτο για αυτή την ετήσια έκθεση. Και εκεί θεωρώ ότι πάρα πολλά θέματα θερμών δικαιωμάτων έχουν να κάνουν για το ότι δεν μπορούμε να προστατεύσουμε αυτούς οι οποίοι παλεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις χώρες. Οπότε αυτό τώρα που θέλω να σας ε, ερωτήσω σχετικά με αυτό και έχω τις εξής ερωτήσεις. Τι νομίζετε, μπορούμε να ξεκινήσουμε μια κοινή προσπάθεια για την ενίσχυση των πολιτικών για να βοηθηθούν αυτοί που παρέχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και έτσι να έχουμε κάποια δράση ε, σε, και έτσι πολλές χώρες να μπορούν να συμμετάσχουν. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε και μέσω των αντιπροσωπιών που δρούν εκτός Ευρώπης αυτά τα σημεία εστίασης ούτως ώστε να μπορούμε να δούμε ακριβώς τι γίνεται με την δράση που αναβάνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι γίνεται με τα άτομα αυτά που παλεύουν για τα δικαιώματα. Νέο μηχανισμό, γιατί όποτε έχουμε αποστολή από το Κοινοβούλιο, συνέχεια τίθεται αυτό το ζήτημα. Όταν πάνε στο εξωτερικό, σε πολλές χώρες. Άρα όλα αυτά μπορούμε να τα συνδυάσουμε και να αναλάβουμε μια κοινή προσπάθεια για τις τρίτες χώρες. Δεν να συμφωνείτε, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα επικεντρώσουμε περισσότερο όσον αφορά το πώς θα προστατεύσουμε τις γυναίκες που μα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και σχετικά με αυτό να δούμε πώς θα συμμετέχουν περισσότερο στο δημόσιο βίο οι γυναίκες και κυρίως όσον αφορά την καταπολέμηση των εξτρεμιστικών ιδεολογικών. Πέστε μου τι πρεσβεύετε. Η Ευχαριστούμε κύριε Παντσέ. Ο κύριος Τόκης. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ. και ευχαριστούμε και τον κύριο Φόρστ. Παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερη προσοχή το έργο του ειδικού εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μάλιστα ε, ξέρω τι, πόσα δεινά υπέστη η Ρουμανία κατά τη διάρκεια του κομμουνισμού και πόσο δύσκολο ήταν να διαμαρτυρηθεί κανείς ή να εξεγερθεί κατά της δικτατορίας. Και χρειάστηκε να αρθεί αυτός, αυτό το τείχος της σιωπής, γιατί ήμασταν φημωμένοι όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι. Γι' αυτό καταλαβαίνω τι μπορεί να περνά ένας ακτιβιστής. Ο κύριος Φόρστ είπε ότι μερικές φορές οι δράσεις μας είναι αντιπαραγωγικές. Γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε συγκεκριμένες ομάδες, αλλά εξαιτία ακριβώς των ενεργειών μας, οι αρχές μας, οι αρχές είναι ακόμη πιο αυστηρές ή πιο αμήλικτες κατά των ακτιβιστών. Πώς μπορούμε λοιπόν να προστατεύσουμε τους ακτιβιστές για να μην μετατραπούν σε αποδιοπομπέους τράγους και να μην ε, υφίστανται συνεχώς επιθέσεις ή στέρηση ελευθερίας ή παράνομες φυλακίσεις. Αυτά τα σημεία πρέπει να επιμένουμε στις, σε αυτά τα σημεία πρέπει να επιμένουμε στις επισκέψεις μας επιτόπου, γιατί για παράδειγμα, στην επίσκεψη στο Βιετνάμ ο εισηγητής δεν μπόρεσε να συναντήσει όλους τους ακτιβιστές που ήθελε. Του απαγορεύτηκε πρόσβαση σε συγκεκριμένες ε, ε, περιοχές ή επαφή με συγκεκριμένους ανθρώπους. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε τους ακτιβιστές και να αναλύσουμε, να προσέξουμε την κατάσταση σε, ιδιαίτερες κρίσιμες, σε ιδιαίτερα κρίσιμες χώρες για να βοηθήσουμε κυρίως ε, εκείνους τους ακτιβιστές. Ο κύριος Γζιμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Φόρστ για την παρουσίαση που μας έκανε. Έχετε πλούσια και προσωπική πείρα στο θέμα των υπερμάχων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις προηγούμενες σας εμπειρίες στο Φόρουμ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε, ε, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο βραβείο Ζαχάροφ που επιβραβεύει ακριβώς την ελευθερία σκέψης μα είναι ιδιαίτερα προσφυλές αυτό το βραβείο, γιατί συνδέεται άμεσα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ε, δημοκρατική μετάβαση. Και από την εμπειρία που είχαμε με την πολύχρονη αυτή απονομή του βραβείου, ε, είδαμε ότι αρχικά ίσως δεν φαίνεται πολύ σημαντικό ότι δίνουμε το βραβείο αυτό στον Α ή το Β αλλά διαπιστώνουμε ότι χάρη στο βραβείο δημιουργείται ένα ολόκληρο κίνημα. Τώρα υπάρχει και ένα ειδικό δίκτυο των βραβευθέντων με το βραβείο Ζαχάροφ. Οπότε είναι σημαντικό αυτό το θέμα και, και το Συμβούλιο επίσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα μπορούσε να συμβάλλει σε ένα τέτοιο δίκτυο, γιατί ένα τέτοιο δίκτυο ακτιβιστών ενισχύει πολύ περισσότερο την, το άκουσμα της φωνής των ακτιβιστών. Ε, μιλήσατε για περιφερειακές διαβουλεύσεις που είχατε και μερικές που επίκυνται. Θα μπορούσατε να μας πείτε ε, ποια περιοχή του κόσμου είναι χειρότερη από την άποψη της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή διαπιστώσατε κάποιες αλλαγές θετικές σε ορισμένες περιοχές. Γιατί φυσικά δεν είναι παντού η ίδια η κατάσταση. Σίγουρα στις χώρες με απολυταρχικό καθεστώς η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Έχουμε γνώση του πράγματος. Αυτή είναι λοιπόν η ερώτησή μου. Επίσης, εμείς επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερως στις ε, σχέσεις μας με τις γειτονικές μας χώρες. Ποια είναι η δική σας ε, αίσθηση για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά τις εξεγέσεις της Αραβικής Άνοιξης γιατί είχαμε και τις τελευταίες εξελίξεις και στις χώρες ανατολικής ε, ε, γειτονίας, αλλά και τα γεγονότα στην ε, Εγγύης Ανατολή. Ποια είναι η δική σας γνώμη. Ευχαριστώ κύριε Ξύπ. Θέλει άλλος κανείς το λόγο. Έχω και εγώ μια σύντομη ερώτηση. Είπατε ότι έχετε προγραμματίσει μια σειρά επισκέψεων. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν ποιο είναι το πρόγραμμά σας και πού θα μεταβείτε μέχρι τα τέλη του έτους. Επίσης μιλήσατε για τις περιφερειακές διαβουλεύσεις. Διαπιστώνετε ε, συγκεκριμένες τάσεις ε, στις επιμέρους περιφέρειες, στην Ασία για παράδειγμα. Είπατε ότι στη συζητήση σας ε, αναφέρετε και την ανάγκη να βελτιωθεί η κατάσταση για τους whistleblowers, αυτούς που καταγγέλουν συγκεκριμένες καταστάσεις. Εμείς διαπιστώσαμε ότι ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό, ούτε στα κράτη-μέλη υπάρχει ακόμη μεγάλη διάκριση μεταξύ ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταγγελόντων. Υπάρχουν εξελίξεις ε, στο θέμα αυτό. Επίσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουμε την δημιουργία προσωρινών καταλυμάτων, ή ε, ασύλων κέντρων υποδοχής για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχετε παραδείγματα βέλτιστων ή χείριστων πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά αυτά τα άσυλα για τους ακτιβιστές. Έχετε αρκετό χρόνο να απαντήσετε. Πρώτα όμως να δώσω το λόγο σε, στην κυρία Μάχελε που είναι εκπρόσωπος μιας τέτοιας οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ που δίνετε το λόγο και στην κοινωνία των πολιτών για να πούμε τα θέματα μας. Καλώς ορίσατε κύριε Φώστ και σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε και οι frontline defenders αναφαντών σα στηρίζουμε. Οπότε με την ευκαιρία να ευχαριστούμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όσα κάνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το ότι αναδεικνύονται συγκεκριμένε περιπτώσει στα ψηφίσματα. Αλλά ευχαριστούμε και την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα όσα κάνουν για την υπόθεσή μα. Ε, Έχουμε την ετησία εκθεσή μας, εδώ έχω κάποια αντίγραφα αν θέλετε και δυστυχώς η αξιολόγησή μας είναι ότι η κατάσταση δεν βελτιώνεται καθόλου όσον αφορά αυτούς που είναι στα στα δικαιώματα. Πάνω από 130 πέθαναν πέρσι, είτε πέθαναν στη φυλακή είτε φωνέθησαν γιατί οι κυβερνήσει κάνουν ό,τι μπορούν για να του εξοντώσουν. Υπάρχουν στρατηγικέ οι οποίε κατά αυτών των αγωνιστών. Φυλάκιση, φόνος, φήμωση με οποιοδήποτε τρόπο. Και όπως είπε και ο κύριος Φως, έχουμε ένα σωρό νομοθεσίες ε, κατασταλτικές, αντιτρομοκρατικοί νόμοι, νόμοι κατά Γενέ πολιτών, κατά της προσβασιμότητας χρηματοδότηση, κατά του διαδηλώνην, κατά της δραστηριότητας των ε, ΛΟΑΔ. Επομένως χρησιμοποιείται το, το δίκαιο, ο νόμος, ούτως ώστε να φημώσει τους ε, αγωνιστές αυτούς και το ένα κράτο ε, αντιγράφει από το άλλο, δανείζεται την νομοθεσία κλπ. Οπότε και εμείς θεωρούμε ότι ενώπιον αυτής της κατάστασης αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η διεθνής κοινότητα στο ανώτατο δυνατό επίπεδο ούτως ώστε να διατεθούν όσο γίνεται περισσότεροι πόροι για να προσταθούν οι αγωνιστές κατά αυτών που προσπαθούν να τους ε, φημώσουν. Επίσης, συχνά εδώ έρχομαι και συζητούμε τι γίνεται για αυτές τις ε, δηλώσει και στην υπηρεσιακή δράση και στο κοινοβούλιο τα λέμε αλλά είδαμε ότι από πλευράς ε, φορέων του επίπεδου πάρα πολύ λίγε δηλώσει υπάρχουν για τους αγωνιστές αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη από αυτέ τι ανακοινώσεις. Καμιά φορά όμως και αυτοί ωφελούνται αν υπάρχει στήριξη ε, δημοσία από αλλού από άλλα κράτη και να γνωρίζει το έργο τους. Και όταν έχουμε τέλος πάντων τέτοιες δηλώσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις, πολλές φορές δεν τους ε, ονομάζουν αγωνιστές. Ε, μιλούμε για πολιτικούς. Τους ονομάζουν ακτιβιστές, bloggers. Αυτό όμως τους αδικεί όσον αφορά το έργο το οποίο επιτελούν και το πόσο σημαντικό είναι για την κοινωνία. Άρα θα πρέπει να τους αγνωρίσουμε. να πούμε τι είναι. Είπαμε για κράτηση, φυλάκιση, υπάγεια στατική διαφόρων χωρών και είπαμε ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαιτεί την αποφυλάκησή τους, την απελευθέρωσή τους. Κύριε Φώστη, είπαμε ότι θα πρέπει χωρίς προϋποθέσεις όλοι αυτοί να ε, βγουν από τη φυλακή, να απελευθερωθούν. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης μας λέει για ε, το ότι θα πρέπει να περνάνε από δίκη. Βέβαια γνωρίζουμε ότι ε, οι δίκες αυτές δεν είναι δίκες, ότι τα, τα δικαστήρια αυτά δεν λειτουργούν ανεξάρτητα. Οπότε γι' αυτό και θα πρέπει να ζητείται η απελευθέρωσή τους. Υπάρχουν κάποιες καλές πολιτικές που μπορούμε να τις ε, ασπαστούμε. Επίσης και το Συμβούλιο Εξωτερικών θα πρέπει να ασχολείται και εκείνο με τους αγωνιστές για να αποδεικνύει πόσο θέμα προτεραιότητας είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό και, στο, και στην ομάδα Κοχόμ και στο πίεση. Κάτι γίνεται, δηλαδή γίνονται αρκετά και αν και ό,τι γίνεται δεν ξέρω, δεν το μαθαίνουμε. Επομένως, έχουμε κάποιες περιπτώσεις, κάποιες περιπτώσεις που έχουν χρονίσει, άρα να, μπορεί να λάβει δραστηριότητα η, η Κόχομ. μιλούμε για κάποιους που είναι πάρα πολύ καιρό στη φυλακή. Παρακαλούμε όλες τις πολιτικές του Κοινοβουλίου να υποστηρίξουν αυτές τις ε, υποθέσεις και τα σχετικά ψηφίσματα. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Να, για το Μπουρούντι, πέντε μέρες μετά το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, κάποιοι άνθρωποι απελευθερώθηκαν. Οπότε παρακαλώ όλες οι πολιτικές ομάδες να στηρίξουν τέτοιες προσπάθειες. Κύριε Φώστερ, μία ερώτηση. Θεωρώ ότι έχουμε κάποια αναδυόμενα κράτη στα Έθνη τα οποία είναι υπέρ των αγωνιστών πέραν των συνήθων υποστηρικτών τους. Τι λέτε, μπορείτε να χτίσετε κάποιες συμμαχίες με αυτά τα καινούργια κράτη, να, όπως η ακτή ελεφαντοστού, που έχουν περάσει νόμους υπέρ αγωνιστών. Άρα, έστω και στο επίπεδο ανακοινώσεων και δηλώσεων, να γίνει κάτι πέραν των συνήθων χωρών που ασχολούνται με τους αγωνιστές. Άρα πέραν των, ε, πέραν των, των, των δηλώσεων δεν πρέπει να γίνει κάτι για τα δικαιώματα αυτών. Τουλάχιστον να γίνει μια ζήμωση, μια συζήτηση σε διεθνές φόρουμ που να αφορά την προστασία τους. Και μέρα μια δεκαετία τέτοιου προβληματισμού κάτι να βγει αυτούς τους αγωνιστές. Έχετε να σου ρωτήσει κύριε τι λέει ο Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλους όσοι έλαβαν τον λόγο. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη, τη σημαντική υποστήριξη που προσφέρει στην εντολή αυτή και σε άλλους από τους συναδέλφους ειδικού συζητητές. Έχουμε όντως ανάγκη να αισθανθούμε πίσω μας το ειδικό βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί και να διατυπώνουμε προτάσεις. Φιλόδοξες μερικές φορές και που δεν είναι αριστές σε ορισμένα κράτη. Ιδιαίτερα εκεί όπου απειλούνται περισσότερο οι αγωνιστές των δικαιωμάτων. Υπάρχουν κάποια κράτη αποφασισμένα. Και είναι δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει προς κάποιες κατευθύνσεις. Για τις κατευθυντήριε γραμμές καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δουλειά που έχει γίνει 10 χρόνια τώρα αφού εορτάσαμε την δεκάτη επέτειο ενός ε, σπουδαίου εργαλείου που δημιουργήθηκε και γέννησε μια δυναμική σε διεθνές επίπεδο που επιτρέπει την ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών. Με χαρά παρακολούθησα τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΑΣΕ, χρήσιμες σε περιοχές, σε χώρες ε, πολύ επιλητικές για τους αγωνιστές ανθρωπινών δικαιωμάτων και με χαρά βλέπω ότι η Ελβετία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και άλλα κράτη ε, σύν το χρόνο να πτήσουν εθνικές κατευθυντήριες γραμμές. Ένα μέσο πολύ χρήσιμο πιστεύω ώστε να αντιληφθούν καλύτερα τα κράτη την ανάγκη να προστατεύουν και οι υπερασπιστές, οι αγωνιστές, ότι έχουν κάποιους που μπορούν, όπου μπορούν να αναζητήσουν άσυλο και προστασία η μη προστασία. Για τις κατευθυντήρες γραμμές Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια και εγώ είχα την ευκαιρία και την τύχη να με υποστηρίξει ε, το Συμβούλιο με τις Περιφερειακές Οργανώσεις. Στις Περιφερειακές ε, Διαβουλεύσεις ζητούσα πάντα να διατυπώνεται το ερώτημα των υπερασπιστών των ανθρωπινών δικαιωμάτων για το πώς αντιλαμβάνονται τις κατευθυντηρίες γραμμές και τη συμπεριφορά των ε, πρεσβειών, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και των κρατών μελών. Όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θα καταγραφεί στην αξιολόγησή μου σε ένα έργο το οποίο θα άξιζε ίσως πιο επιστημονική προσέγγιση, αλλά πάντως θα συμπληρώσει την πρώτη αξιολόγηση των ε, ορισμένων κρατών από το Κοινοβούλιο. Οι κατευθυντήριες γραμμές καταρχάς είναι γνωστές, από τους, είναι γνωστές τους ε, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ξέρουν που πρέπει να στραφούν. Αλλά δυστυχώς δεν είναι δυνατόν αυτό σε όλες τις χώρες και χωρίς να θέλω από τα δύο παραδείγματα που θα σας αναφέρω να πω ότι είναι χαρακτηριστικά και των λοιπών κρατών, θα σημειώσω ότι δεν ισχύει πάντα αυτό. Πρώτο παράδειγμα λοιπόν, η πρώτη μου αποστολή, κυρία Πρόεδρε, ήταν στο Μπουρούντι για 15 μέρες, σε δύσκολη περίοδο πριν από εκλογές, όπου διατυπώνονται σαφείς απειλές κατά των υπερασπιστών των ανθρωπινών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα ενός που ε, κατήγγειλε τη βούληση του ε, Προέδρου του Μπουρούντι να ε, είναι υποψήφιος για τρίτη φορά και την ε, άρνησή του να εγκαταλείψει την εξουσία. Ε, αυτό ισοδυναμούσε για τον Μπουρούντι με έγκλημα καθοσιώσεως, φυλακίστηκε, απειλήθηκε και κινδυνεύει και η ζωή του ακόμη. Στην επίσκεψή μου λοιπόν στον Μπουρούντι φυσικά στράφηκα στην ε, πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τη ζητήσω την, υλοποίηση, την ενεργοποίηση του μηχανισμού που προβλέπεται, δηλαδή του ταμείου που προβλέπεται για να του εξασφαλιστεί άσυλο, διαφυγή από τη χώρα, άσυλο στον ίδιο για να μπορέσει να φύγει από το Μπουρούντι. Αυτό η γυναίκα του που ήταν έγκυο στα δύο παιδιά του. Το, το κύριο δεδομένο των απειλών που είχαν εκτοξευθεί εναντίον αυτού του ανθρώπου ήταν να εξασφαλίσουμε τη ε, διαφυγή του από τη χώρα. Δυστυχώ όταν στράφηκα εγώ στην ε, πρεσβεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είχε ενεργοποιηθεί ακόμη ο μηχανισμό, άρα έπρεπε να καθυστερήσει η διαδικασία μέχρι ότου ε, αναπτυχθεί το ερωτηματολόγιο από την Πρεσβεία για να δει εάν ε, αν πληρούσε τις προϋποθέσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάστηκε να περάσει πολλή χρόνος και με αρκετές δυσκολίες μόνο μπόρεσε να ε, βρεθεί ασφαλές καταφύγιο για τον άνθρωπο αυτό και την οικογένειά του. Χρειάζεται λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις να γίνει η κατάρτιση, η παιδαγωγική αυτή δουλειά που χρειάζεται και η εργαλειοθήκη εντό εισαγωγικών, το toolkit που θα πρέπει να έχουν στη θέση του έτοιμο οι υπηρεσίε για να μπορούν να ανταποκρίνονται ε, καθυστέρηση στις κατευθυντήριες γραμμές και τις προποθέσει τους. Ένα άλλο παράδειγμα από την Μπογκοτά. Η Κολομβία, όπω ξέρετε, είναι ένα κράτο το οποίο έχει εκτοξεύσει πολύ ε, άμεσες και βίες ε, απειλές κατά των αγώνων των ανθρωπινών δικαιωμάτων και σε μια τέτοια διάσκεψη στην Κολομβία, στην Πογκοτά, ακούσαμε ένα νομικό να, λέει, να μου λέει μάλλον, στη διάσκεψη, Κάθε μέρα φωνεύεται και από ένα ε, αγωνιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάθε μέρα, 55 του προηγούμενου χρόνου αντιστοιχούν σε ένα θάνατο την ημέρα. Ένα ζήτημα λοιπόν το οποίο θίξαμε στις επαφές μας με την ε, Πρεσβεία και ζήτησα από την Ορβηγία να οργανώσει μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση μια ε, συνεδρίαση των πρεσβευτών των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να συζητήσουμε την υλοποίηση των, την ενεργοποίηση των κατευθυντικών γραμμών για την Κολομβία. Δουλειά γίνεται. Εκεί είναι γνωστό ο μηχανισμό. Οι υπερασπιστέ των ανθρώπινων δικαιωμάτων γνωρίζουν το μηχανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά καλά, είναι ενήμεροι. Αλλά υπάρχουν προβλήματα ίσω πολιτική φύση, τα οποία θα ξαναεπαληθευθούν και την μπορεί να επαναληφθούν και σε άλλε χώρε. Υπάρχει ένα σημαντικός μηχανισμός λοιπόν εθνικής προστασίας των ε, αγωνιστών, 180 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο δαπανά η Κολομβία για την προστασία τους, για τους σωματοφύλακες, τα τεθωρακισμένα αυτοκίνητα, την φύλαξη των κτηρίων ε, και των οικογενειών των αγωνιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απειλούνται. Άρα είναι σημαντική η επένδυση. Αλλά πολλοί από αυτού, του αγωνιστέ δεν τολμούν να στραφούν στο μηχανισμό τη Κολομβία. Γιατί, Γιατί η Κολομβία έχει δώσει ως υπεργολαβία το έργο αυτό της φύλαξη σε ιδιωτικέ εταιρείε φύλαξη, για τις οποίες οι αγωνιστές μου λένε ότι οι ίδιες ήταν οι αυτούργοι των παραβιάσεων των δικαιωμάτων στο παρελθόν. Δεν μπορούν λοιπόν να αισθανθούν ασφαλείς στα χέρια αυτών που ήταν οι αυτούργοι των παραβιάσεων των δικαιωμάτων στο παρελθόν στην ίδια χώρα. Άλλο ενδιαφέρον για την Κολομβία, όταν απευθύνθηκα στον πρεσβευτή σας, τον πρεσβή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ρωτήσω γιατί δεν αξιοποιείται το ταμείο που αφορά την επανεγκατάσταση αγωνιστών των, των ανθρωπινών δικαιωμάτων, η απάντηση που πήρα ήταν τα τελευταία δύο χρόνια την έχουμε, το έχουμε αξιοποιήσει το ταμείο αυτό τρεις φορές. Ωστόσο, Φοβούμαστε ότι εάν αξιοποιηθεί πολλές φορές αυτό το ταμείο για να διαφύγει στο εξωτερικό ένας αγωνιστής, θα δώσουμε την εντύπωση στην κολομβιανή κυβέρνηση ότι δεν τους εμπιστευόμεθα στην, ε, στο καθήκον αυτό που έχουν να προστατεύουν. Δηλαδή και ο αγωνιστής των πρώτων δικαιωμάτων φοβάται να, καταφύγει, να προσφύγει στον εθνικό μηχανισμό γιατί ο, η υπηρεσία φύλαξης ε, η τωρινή είναι ο δίμιος του παρελθόντος και από την άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια αισθάνεται μια μηχανία λέγοντας ότι εάν ε, προσφέρει προστασία στους αγωνιστές αποστέλει μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν είναι ικανή να τους προστατέψει η ίδια, άρα πρέπει σε πολιτικό επίπεδο να βρεθεί μια διαφορετική λύση. Για τις γυναίκες αγωνιστές των ανθρωπινών δικαιωμάτων έχω μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Ύστερα από την οργάνωση κατόπιν προτάσεως της ε, Ένωση Γυναικών ε, που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια σειρά από επαφών μόνο με γυναίκες. Είχα ζητήσει δηλαδή από του άντρες να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Υπήρχαν γυναίκες δηλαδή που μου έλεγαν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε μπροστά σε άντρες συναδέλφους. Και όντω, είδα να αναπτύσσεται μια νέα δυναμική στη σχέση μεταξύ γυναικών αγωνιστριών και του υποφαινομένου που είχα πάει για να τις ακούσω. Μου είπαν πράγματα που δεν είχαν υποθεί παρουσία των αντρών ε, συναδέλφων τους για ιδιαίτερα προβλήματα, απειλές, ε, παρενόχληση, ε, κινδύνους και βέβαια όσον αφορά την ε, σεξουαλική παρενόχληση και απειλές είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και στις αραβικές χώρες και στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική μια στρέβλωση της εικόνας απειλές μέσω του Twitter, μέσω των ε, λογαριασμών ε, Facebook, ε, μέσω υφαρπαγής των προσωπικών του στοιχείων και παρουσία φεριπίν στην σελίδα τους, του προσώπου τους με το σώμα μιας άλλης γυναίκας γυμνό που βέβαια ντροπιάζει και τις ίδιες και, την και τις οικογένειές τους. οι άντρες συναδελφοί τους δεν τους αφήνουν επαρκή χώρο, έχουν ε, σοβινιστική στάση απέναντί τους. Άρα για τις γυναίκες που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα πολύ δουλειά μένει να γίνει ακόμα, όχι μόνο από τη διεθνή κοινότητα, αλλά και από τις ε, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις της ίδιας που πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο θεώρησης των γυναικών που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την προστασία της ασφάλειας και την ασφάλεια των ε, υπερασπιστών. Έχει γίνει λόγος για shelter cities, πόλεις άσυλα. Χαιρετίζω εδώ τις προσπάθειες των ε, κάτω χωρών που προσφέρουν ασφαλές καταφύγιο για τρεις μήνες εκείνους που απειλούνται από ιδιαίτερα σοβαρές απειλές και τους προσφέρει κατά την ε, υποδοχή ψυχολογική υποστήριξη, γλωσσική κατάρτιση ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν και να γυρίσουν να αγωνίζονται στη χώρα τους όταν έρθει η ώρα. Στη Γενέβη την προηγούμενη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με πολλούς πρέσβες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το μηχανισμό αυτών των πόλεων καταφυγίων. Ο πρέσβης της Αυστραλίας, σε παραδείγματι, μου είπε ότι για την, περιφέρεια, για την περιοχή της Ασίας τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αυτές οι λύσεις, αλλά φοβάται ότι μπορεί αυτό να αποτελέσει πόλο έλξης για πολλούς ε, που θα έρθουν να στήσουν άσυλο στην ε, Αυστραλία. Δηλαδή, λέει, δεν θέλω να έρχονται και να ζητούν άσυλο μόνο και μόνο γι' αυτό. Και άλλοι εκπρόσωποι και από άλλε χώρε και από άλλε υπήρου ε, έθιξαν το θέμα αυτό, λέγοντα ότι ίσω στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Λατινική Αμερική θα ήταν σκόπιμο να απτυχθούν τέτοιου είδου πόλει άσυλα. Και δεν αντιλαμβάνονταν πολλοί πρέσβει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πρόσφυγες, δεν ζητούν άσυλο ότι πάνω απ' όλα του ενδιαφέρει άπαξ και περάσει ο άμεσο κίνδυνο να γυρίσουν στι χώρε του για να συνεχίσουν να αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήρθα σε επαφή με του Ολλανδού ε, συναδέλφου που με ενημέρωσαν ότι από τη στιγμή που εγκαθιδρύθηκε το σύστημα και άρχισε να λειτουργεί, δύο μόνο από αυτού που είχαν βρει ε, ασφαλέ καταφύγιο ζήτησαν στη συνέχεια άσυλο, μόνο και μόνο γιατί ήταν πολύ οξύες και άμεσες οι απειλές εις βάρος τους. Ε, όλοι οι υπόλοιποι που είχαν αναζητήσει καταφύγιο στις πόλεις αυτές δεν ε, μετατράπηκαν σε πρόσφυγες, δεν ζήτησαν μετά άσυλο και πρέπει να γίνεται πάντα η διαφοροποίηση. Την επόμενη εβδομάδα στη Γενέβη με το Συμβούλιο Εθνών Δικαιωμάτων, ε, με προεδρία του Ολλανδού ε, πρέσβη θα γίνει συζήτηση σε πάνελ όπου νομίζω θα μπορέσουμε να συζητήσουμε διεξοδικά τι είναι αυτές οι πόλεις καταφύγια. Εάν μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβάλλει τις ιδέες αυτές μέσα στο ίδιο το Κοινοβούλιο αλλά και σε σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια για να εμπλακούν στη συζήτηση για το θέμα αυτό σε εθνικό επίπεδο, να υπάρξει η ιδέα της ανάπτυξης των πόλεων ασύλου και τη δυνατότητα παροχή ασφαλού καταφυγίου για τρει μήνε τουλάχιστον για του ανθρώπου αυτού που θα μπορέσουν στη συνέχεια όταν είναι πιο ασφαλείς να επανέλθουν στη χώρα τους, να ξαναοργανωθούν, να αποκαταστήσουν την, ε, το, έργο τους και τις συνδέσεις τους και να ξαναρχίσουν τη δουλειά. Για τις χώρες έχω ένα χρονοδιάγραμμα επισκέψεων που, που με δυσκολία πολλές φορές μπορώ να τηρήσω. Έχω χώρες που καλούνται, που με προσκαλούν μένα αλλά μου διαθέτουν τόσο περιορισμένο ε, χρόνο που δεν ε, υπάρχει ουσία. Για την ε, Τουρκία, παραδείγματι, χαρακτηριστικά έχω αποδοχή της επίσκεψης πέντε μέρες μόνο, όσο δίνουν στους ειδικούς ε, εισηγητέ. Εμένα σκοπό μου να μην περιοριστώ στην πρωτεύουσα, αλλά να φτάσω μέχρι τα σύνορα της Συρίας, να κοιτάξω τους πιο απομακρυσμένου πληθυσμού, του πιο απομονωμένου πολίτε και να δω στην περιοχή αυτή την πιο επικίνδυνη το πώ μπορεί να ε, βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπους, ιδιαίτερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περιμένω να με στηρίξει αν υπάρχει τρόπος ε, στην επίσκεψη αυτή. Για το Κυργιστάν υπάρχει μια, ένα αίτημα για επίσκεψη που δεν θα γίνει δεκτό κατά πάσα πιθανότητα στην ε, Ρωσική Ομοσπονδία, στη Λευκορωσία, στο Μεξικό. Στις Φιλιππίνες που ελπίζω ότι θα μπορέσω να πάρω τη σχετική άδεια προς το τέλη του έτους την Αφρική, Φερρυπίν Κένια, Ζιμπάμπουε, άλλες αφρικανικές χώρες για τις οποίες έχω ζητήσει την άδεια να επισκεφθώ και θα ήθελα ή μη τι άλλο να αισθάνομαι ότι πίσω μου έχω το, το βάρος, το ειδικό βάρος των κρατών μελών, των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν δεν λαμβάνω τη σχετική άδεια, να πάω επισήμως δηλαδή σε επίσκεψη σε μια χώρα, έχω προτείνει την αξιοποίηση ενός ε, μηχανισμού παραδρομής, δηλαδή ζητώ να με προσκαλούν οι πρεσβείες, οι πρεσβείες σας. Να πάω στη χώρα για να συμμετάσχω σε ένα συνέδριο, σε ένα πάνελ, σε μια συζήτηση. Κάποιες από αυτές τις πρεσβείες με έχουν προσκαλέσει σε χώρες δύσκολες, περίπλοκες, για τις οποίες δεν θα έπαιρνα άδεια να επισκεφθώ. Αλλά κατόπιν προσκλήσεως μιας πρεσβείας μπορώ να μεταβώ στη χώρα. Ενημερώνω τη μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας στη Γενέβη ότι θα μεταβώ. Δηλώνω ότι δεν πρόκειται να προβώ σε δημόσιες δηλώσεις ή ανακοινώσεις στο Twitter κτλ. Πάω μόνο για να συναντηθώ με αγωνιστές των ανθρωπινών δικαιωμάτων, με ακτιβιστές και πάντα μετά από αυτές τις συνεδριάσεις φροντίζω να αφήσω μισή ή μία μέρα ολόκληρη άδεια ώστε να έχω επαφές σε επίσημο επίπεδο, όχι ανώτατο, όχι υπουργού δηλαδή, αλλά ε, διευθυντές, γενικούς διευθυντές από τα Υπουργεία στα θέματα τα πολιτικά των εσωτερικών, των κοινωνικών υποθέσεων, ώστε να συζητήσουμε θέματα ουσίας που έχουν να κάνουν με τους αγωνιστές αυτούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν μπορούσατε να με στηρίξετε σε αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο. Πολλοί ακτιβιστές επίσης έχουν έρθει να επισκεφθούν εμένα. Έχω ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα επισκέψεων μετά από, τις, ε, μετά από τα αιτήματα των ε, ε, των αγωνιστών αυτών. Προπολογισμό από τα Ηνωμένα Έθνη επιπλέον δεν έχω, άρα έχω και οικονομικό περιορισμό. Η Νορβηγία όμως με έχει στηρίξει οικονομικά που έχει ηγηθεί αυτής της πρωτοβουλίας και μου έχει επιτρέψει χάρη σε, σε προσκλήσει από την κοινωνία των πολιτών να έρθω σε επαφή με τους ακτιβιστές ε, οι οποίοι μου λένε πάντα θέλουμε να είστε παρόντες επί τόπου, θέλουμε να είστε αυτοί οι οποίοι, όπως λένε στα αγγλικά, θα voice our concern, θα μεταφέρεται, θα καταστεί τα φερέφωνα των μελημάτων μας. Ε, δεν μπορούν όλοι τους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, δεν μπορούν όλοι τους να έρθουν μέχρι την Ευρώπη ή το Συμβούλιο των Ανθρωπινών Δικαιωμάτων, δεν μπορούν όλοι τους να φτάσουν μέχρι τη Γενική Συνέλευση. Πρέπει να είναι στο πλευρό τους ο εισηγητής να έρχεται να τους βλέπει και να μπορεί να μεταφέρει στον έξω κόσμο τις ανησυχίες τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για τους λεγόμενους whistleblowers, αυτούς που καταγγέλουν κακό κείμενα. Σας έχει απασχολήσει και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ξέρω. Είχαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντικές τέτοιες καταγγελίες. Υπάρχουν μικρότεροι βεληνικούς καταγγελίες που όμως χρήζουν καλύτερης προστασίας. Γι' αυτό θα δείτε στην έκθεσή μου ότι έχω δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα στο θέμα αυτό και σε συνεργασία. Και έχω έρθει πολύ κοντά στον συνάδελφο David Kay που είναι ο ειδικό ηγετής για την ελευθερία της έκφρασης προκειμένου να υπάρχει μια κοινή έκθεση για τις απειλές ε, που επικρέμονται από αυτών των ε, καταγγελόντων, οι οποίες δεν προέρχονται πάντοτε από κρατικές δομές, αλλά από υπερεθνικές, πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες πολλές φορές διαθέτουν τα στοιχεία των, μεταβιβάζουν τα στοιχεία των ε, καταγγελόντων αυτών σε κρατικές δομές. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ελπίζω στην επόμενη αυτή έκθεση που σκοπεύω μαζί με τον κύριο Κέι να διατυπώσουμε, να είμαστε θέση να εκφράσουμε και υποδείξεις προς κράτη, προς εθνικές δομές ανθρώπινων δικαιωμάτων, προς την κοινωνία των πολιτών, αλλά και προς υπερεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες όπως ξέρετε και λόγω των δικτών που έχουμε υιοθετήσει τα Ηνωμένα Έθνη για το ρόλο και την ε, ε, συνυπευθυνότητα των μεγάλων υπερεθνικών επιχειρήσεων στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικές. Κοιτάω λίγο στι ε, σημειώσεις μου αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο έχω λησμονήσει. Η σύμβαση. Η ερώτηση τη Frontline για τη σύμβαση. δεν έχω απάντηση προ το παρόν. Έχουμε αναπτύξει μια σειρά από πρότυπα σε διεθνές επίπεδο, συμβάσεις έχουν αναπτυχθεί και όταν κοιτάμε το ποσοστό υλοποίησης των συστάσεων από τα όργανα της συνθήκης, ε, θέλω να πω ότι ανησυχούμε για τον πολύ περιορισμένο βαθμό συνεργασίας των κρατών. Διαβούλευση για μια σύμβαση τουλάχιστον θα σήμαινε ότι τα κράτη-μέλη κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι, έστω και αυτά που δεν είναι οι καλύτεροι ε, σύμμαχοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κάτσουν να ακούσουν, έστω και αν δεν τους αρέσει, ε, προτάσεις και θέσεις. Ίσως έτσι μπορούμε να αντιδράσουμε στις, ε, στην ε, αρνητική του στάση εναντί των αγωνιστών. Επίσης, τα διάφορα βραβεία οι κάτω χώρε έχουν το βραβείο τη Τουλίπα. Το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίση ένα ε, βραβείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, η Γαλλία επίση. Ε, είναι ένας καλός τρόπος να επιβραβευθούν και να προβληθούν αυτοί οι αγωνιστές. Πολλέ φορέ όμως προβάλλονται τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα και λησμονούνται αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται στη μικρή κλίμακα, στι πιο απομακρυσμένε περιοχέ που έχουν πιο πολλού κινδύνου και που χρειάζονται πιο πολλή προστασία επίση. Γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να φτάσω μέχρι κάθε άκρη για να συναντηθώ μαζί του, να του δώσω φωνή και να μεταφέρω τα λόγια αυτών των ανθρώπων των οποίων η φωνή δεν ακούγεται συχνά. Πρόεδρε, νομίζω ότι έχω απαντήσει σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις και αν δεν το έπραξα ζητώ συγγνώμη. Μερικές φορές τις σημειώσεις μου ε, δεν ε, είναι δυνατόν να αποκρυπτογραφηθούν. Σας ευχαριστώ. Εκτενέστατες οι απαντήσεις σας. Και επειδή θέσαμε ερωτήσεις και για συγκεκριμένες χώρες ή περιφέρειες, φαντάζομαι στην ε, η δική σα έκθεση που υπάρχει στο διαδίκτυο μπορούμε να βρούμε περισσότερε λεπτομέρειε. Έχουμε δύο εκθέσει. Καταρχήν την ετήσια έκθεση που υποβάλλουμε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εκεί παρουσιάζω το όραμα τη θητεία μου και τι βασικέ προτεραιότητε τη θητεία μου. Πώ θα δουλέψω δηλαδή και μετά από τρία χρόνια θα κάνω μια αξιολόγηση τη εφαρμογή των προτεραιοτήτων μου και θα ενημερώσω τα κράτη-μέλη για την επόμενη τριετία ευελπιστώ να ανανεωθεί η θητεία μου. Επίσης έχουμε την έκθεση με τις ανακοινώσεις της πληροφορίες που έχω λάβει από οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών ή από θύματα με τις απαντήσεις που έχουν δώσει οι ενδιαφερόμενες χώρες. Οπότε μπορείτε να κάνετε κλικ και σε απαντήσεις των κυβερνήσεων και στις ε, καταγγελίες που έχουν γίνει. Βλέπετε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση των χωρών, σε ό,τι αφορά τις συστάσεις μου ή τις υποδείξεις με βάση συγκεκριμένε υποθέσεις. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε την πρωινή μας συνεδρίαση. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Είχαμε μεγάλη ε, χαρά γι' αυτό και καλή σας τύχη στην ε, επόμενη σας συνεδρίαση με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εμείς θα συνεχίσουμε το απόγευμα στις 3 με το διευρυμένο Προεδρείο και κατόπιν ε, θα έχουμε μονόρι ε, συνεδρίαση με εκπρόσωπο της ΥΠΑ της Αρμοστίας με ειδικό θέμα την κατάσταση των σύρων προσφύγων στο Λίβανο. Καλό σας μεσημέρι.